much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Right. Um, good afternoon, everybody. Σας καλωσορίζω όλους. Γνωρίζω ότι δεν είμαστε όλοι εδώ, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί ε, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μας προειδοποιούν γι' αυτό. Is, uh, number 10, uh, which is the vote on... Λοιπόν, το 10, η ψηφοφορία Κλίντς. Εφόσον έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας, παρακαλώ μπορούμε να τις ελέγξουμε. Ξέρω ότι ο Σβέν δεν έχει την δική του κάρτα. Ο Πιτέλα δεν έχει ούτε αυτό στη δική του. Παρακαλώ. Τεστ με τις κάρτες παρακαλώ. Ψηφίζετε δοκιμαστικά. We're having a secret ballot. Yeah, secret ballot on do you like the person sitting next. Ναι, θα κάνουμε μυστική ψηφοφορία για το αν σας αρέσει ο παρακαθήμενός σας. Right. Okay. So, so, so we've got three missing now. We've got... Λοιπόν, τρεις λείπουν, ένας σοσιαλιστής, ένας πράσινος Λοιπόν, δοκιμάστε να ψηφίσετε δύο φορές. No, we can tell. It says 64 and 65. <laughs> Same person. It, it, it works if you're in different rooms, but oh well. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει κάποιος πήγε να ψηφίσει αστειευόμενος ε, δύο φορές με την ίδια κάρτα σε δύο διαφορετικές θήκες. Okay, I'll be ready then. Then, um, first of all, compromise C. All Λοιπόν, συμβιβαστική C αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 47 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 48 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική D αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 52 και 53 μαζί ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές 54 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτονται θα υπάρξει έλεγχος για την 54 παρακαλώ And okay, the vote's closed and there's one extra in but it's still lost by one. Λοιπόν, ε, λείπει μία ψήφος ε, δεν, ε, για να περάσει απερίφθη. 56 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 57 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ γιατί 57 δεν είναι καθαρό. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Δεν έχει σημασία ένας-δύο αν δεν ψήφισαν γιατί υπάρχουν 20 κατά και 13 υπέρ. Λοιπόν, περνώ τώρα στην 58. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 60 καταπίπτει, περνάμε στην 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική ή αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτό. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική F α όχι ξανά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 64 ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται Συμβιβαστική F κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η Τζούρι 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική I αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβιβαστικό J υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβιβαστικό K υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβιβαστικό L αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτό η 109 τώρα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 109 Has everybody voted? Votes. Ψηφίσατε όλοι. Απερίφθη. Α, πρέπει να προσθέσουμε και κάποιους. Είναι ισοπαλία λέει η πρόεδρος. Κύριος Πιτέλα. Πώς ψηφίζεται κύριε Πιτέλα. Υπέρ. Οπότε είναι 16 υπέρ και γίνεται δεκτή. Εκατόν εννέα δεκτή λοιπόν. Η εκατόν δέκα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και εδώ παρακαλώ στην 110 ψηφίζουμε την 110 Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες σας. Hm, hm, hm. Ορμήστε λέει η πρόεδρος. Έχουμε άλλους δύο με δυνατότητες ψηφοφορίας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πιέστε παρακαλώ τα κουμπιά σας. Λοιπόν, τώρα ψήφισαν όλοι. Ευχαριστώ. Και απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τζούρι 2 δεύτερο τμήμα υπέρ Το δεύτερο τμήμα λοιπόν της Τζούρι 2 ψηφίζουμε πρώτα το πρώτο τμήμα λέει το η υπέρ το πρώτο τμήμα κατά Αποχές. Δεκτό το πρώτο. Τώρα το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 και 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβιβαστικό M αγγλικό. Α, όχι. Πρώτα το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τώρα συμβιβαστικό M αγγλικό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική τώρα ένα Αγγλικά σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Πηγαίνουμε τώρα στην 119 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή 119, 122 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή 122. 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή 124 υπέρ κατά αποχές εν πάση ηλεκτρονικός έλεγχος για την 124 δεν ήταν καθαρό ψηφίσατε όλοι παρακαλώ πέρα της ψηφοφορίας δεκτό και άλλοι δύο κατά. 20 με 20 λοιπόν. Συνεπώς καταπίπτει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην 125. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Συμβιβαστική. ου αγγλικά υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή 128 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική πία γλυκό υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές δεκτή 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές δεκτή 147 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 147 παρακαλώ λοιπόν ψηφίσατε όλοι απερίφθη 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή 149 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 150 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 150 ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορίας δεκτή 151 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Λοιπόν, τζούρι 6, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 158. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Α, για μια στιγμή. Κάποιος έχει δει το λόγο. Λοιπόν, θα, θα, θα ακυρωθεί η προηγούμενη ψηφοφορία και θα ξαναγίνει η ψηφοφορία για την 158 παρακαλώ Αρχίζουμε πάλι για την 158. 158. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 159 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 160 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη 161 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 162 υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή 165 υπέρ κατά αποχές απερίφθη αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβιβαστική R αγγλικά υπέρ κατά αποχές δεκτή 173 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 170 α όχι ηλεκτρονικός έλεγχος για την 173 Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Λοιπόν, πόσες επιπλέον ψήφους έχουμε λοιπόν. Απερίφθη. Λοιπόν, 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 176 υπέρ κατά αποχές δεκτή 177 υπέρ κατά αποχές για την 177 ηλεκτρονική ψήφος όχι υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική S αγγλική σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα δεκτή δεύτερο υπέρ κατά το δεύτερο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 187. Θέλετε να υπάρξει έλεγχος ηλεκτρονικός για την 186. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 187 υπέρ. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ψηφίζει μόνο ο Βόλφ μόνος του. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 188 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 189 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 189. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη με τρεις ψήφους συν μία ψήφος του Διώγου και άλλη μία ψήφος. Ο κύριος Πιτέλα έχει πλέον την κάρτα του. Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα καταπίπτει, τι γίνεται. Α, τότε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 189 μόνο του. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Περνώ στην 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 91 υπέρ. κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 3 υπέρ κατά ξαναρχίζω την 3 κατά αποχές απερίφθη τέσσερα υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 4 Πέρας ψηφοφορίας έχουμε δύο που πρέπει να ψηφιστούν, να προσθεθούν έτσι, δεν έχουμε τίποτα να αφαιρεθεί. Εγκρίθηκε λοιπόν με μια ψήφο διαφορά. 19 συν 21 υπέρ, 20 εναντίον. Εγκρίθηκε. Και πάμε στην τροπολογία 6 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 7 υπέρ. Καταπίπτει λέγεται. Όχι, λέει ότι είναι συμβατή. και 7 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 8 υπέρ κατά αποχές νομίζω αυτή απορρίφθηκε αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 8 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλες και όλοι πράγματι απορρίφθηκε λοιπόν αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 10 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το πρώτο δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Jury C υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 28 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στο συμβιβασμό Β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 38 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Και τώρα με τις κάρτες θα ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Σαφώς εγκρίθηκε. 27 υπέρ, 14 αποχές. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε ποιοι ευρωβουλευτές ψηφίζουν και δεν έχουν κάρτες, ώστε να ξέρουν οι υπόλοιποι. Σβέν Γκίγκολτ και Διόγκο Φέο. Ο κύριος Πιτέλα Αρχικά δεν είχε, αλλά τώρα έχει την κάρτα του εντωμεταξύ. Αυτά. Okay. Εντάξει. Και περνάμε τώρα, συνεχίζουμε. Έχουμε αλλαγή σε σχέση με την γραμματεία. Εντάξει, αλλά θα συνεχίσω ούτως ή άλλως. Πρόκειται για την έκθεση <clears throat> Ashley Fox ε, για την εταιρική διακυβέρνηση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Όλοι έτοιμοι για την ψηφοφορία, εντάξει. Παράγραφος 1, αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ήμκο 1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ήμκο 3, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ήμκο 5, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Πολύ φασαρία. Ησυχία παρακαλώ. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός β, τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμό Γ, σι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. συμβιβασμό Δ, D, πώς είπατε, χωρί μικρόφωνο η παρέμβαση. Α πάμε στην τροπολογία 14 λέγεται. Α, μάλιστα, καταπίπτει η ΔΕΛΤΑ και πάμε στην τροπολογία 14 τώρα, μάλιστα, που είναι αρκετά παρακάτω στην επόμενη σελίδα. Η δική μου τροπολογία, τροπολογία 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός ή ε, όχι, αυτή στιγμή πρέπει πρώτα να κάνουμε την 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός ε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 22 υπέρ κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ήμκο 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 29 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε την 30. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αν επιθυμείτε. Ήταν σαφές για μένα. Η 30 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 30. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας λοιπόν. Τελειώνει η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. Κύριε Φέο, τι γίνεται. Διέγκο Φέο. Ευχαριστώ, εντάξει. So it's carried. Εγκρίθηκε λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Right. Right. Not to be... Πολύ καλά. Έχουμε την τροπολογία 32 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τώρα, jury, 7, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τζούρι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ως προσθήκη Τζούρι 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τζούρι 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τοπολογία 36 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Τζούρι 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Τζούρι και εγώ, Sharon Bowles, υπέρ λοιπόν, κατά χωρίς αριθμό. Αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 14. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τζούρι. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Αποσύρθηκε αυτή. Τα υπόλοιπε καταπίπτουν. Ήμκο 14 η επόμενη νομίζω. Εντάξει, σωστό. Καταπίπτει η ΙΜΚΟ. Έχουμε την τροπολογία 43 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε. Να ξαναδοκιμάσουμε. Η 43 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Τζούρι 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. ΙΜΚΟ 10 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. ΙΜΚΟ 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Σαφώς εγκρίθηκε. Συμβασμός G υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτουν οι υπόλοιπες. Jury 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός H μια στιγμή συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Jury 2 δεν θα ψηφιστεί εντάξει η 60 θα ψηφιστεί η 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 61 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 62 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αυτή τώρα jury 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τζούρι 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Η 64 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την Τζούρι 3. Εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας, τέλος ψηφοφορίας και εγκρίθηκε μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. hang on. Sorry about this. Wrong phone. Go away. <laughs> um, we're now on 64. 64 λοιπόν. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 65 υπέρ. Κατά αποχές 65 ξαναψηφίζουμε. Σηκώστε τα χέρια σας. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός. Άι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 69 λέει τώρα. 69 δεν την έχω βρει ακόμα. Εντάξει, 69 λοιπόν. Υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Πού πάμε τώρα. Απολογία 70. No, 70 is to be voted as well. Και η 70 θα ψηφιστεί. Η 70 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τώρα συμβιβασμός J υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Where do we go to now? Και πού πάμε τώρα. Ήμκο 19, μάλιστα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 11 υπέρ. Κατά. Ήμκο 11 ξανά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τζούρι 11. Δεν έχει ψηφίσει, δεν ψηφίζεται. Τζούρι 22. Τζούρι 11 είναι δική τους αρμοδιότητα. Τζουρ 22 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 78 υπέρ, κατά, Δεν ξέρω πώς ψήφισαν οι σοσιαλιστές. Έστω, εντάξει, εγκρίθηκε αυτή. 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Τζούρι 11, δεν θα ψηφιστεί. Ήμκο 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 80 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 81 υπέρ, κατά αποχές ε, δεκτεί αυτή. Ήμκο 4 την ψηφίσουμε. Όχι, καταπίπτει. Ήμκο 13 λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Αρχικό κείμενο καταπίπτει. 82 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε εδώ. Είναι το πιο εύκολο. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 82. Ψηφίσατε όλοι. εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. Με δύο ψήφους διαφορά. Με μία, εντάξει, με μία ψήφο διαφορά εγκρίθηκε. 83 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 85 υπέρ, κατά, αποχές Καταπίπτει λέγεται στην πρόεδρο. Μάλιστα καταπίπτει. 87 λοιπόν. 87 υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. 88 υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. 89 υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Κάποιος ζήτησε να, κάνει, να γίνει κάτι. Τι λέτε. Ποια είναι αυτή που ζητάτε. Χωρίς μικρόφωνο. Την 89. Θα ελέγξουμε την 89. Πολύ καλά λοιπόν. Όλα εντάξει. Απορρίφθηκε πράγματι λοιπόν, βλέπετε. Λοιπόν, Τζούρι 23 δεν θα ψηφιστεί. Και πάμε στην ΙΜΚΟ 17, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. ΙΜΚΟ 7, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αυτή. Τζούρι 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τζούρι 24 δεν θα ψηφιστεί. Η 95 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφορίας. Μάλιστα, τι βλέπουμε εδώ. Ένας πάνω ή ένας κάτω, καταπίπτει ούτως ή ας καταψηφίστηκε. 96 υπέρ, κατά. Δεν βλέπω να σηκώνετε τα χέρια σας. Παρακαλώ μεγαλύτερη συμμετοχή. 96 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίφθηκε. 97 υπέρ, κατά. Αποχές, θα ελέγξουμε την 97. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Απορρίφθηκε λοιπόν. Μάλιστα. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 100 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε 101 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 102 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 103 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ την 103 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Εγκρίθηκε λοιπόν, μάλιστα. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Η 105 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 109 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 110 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός και κάπα υπέρ κατά αποχές. Να ξαναψηφίσουμε αν θέλετε το K συμβιβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 114 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 115 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τζούρι 26 δεν θα ψηφιστεί 116 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 117 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός L υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην 120 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 120. Ψηφίσατε όλοι. Δύο από εσά δεν ψήφισαν, αλλά έστω τέλος ψηφοφορίας καταψηφίστηκε. Ακόμα και αν είσαστε εσείς υπέρ Σβέν, πάλι καταψηφίστηκε. Η 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός εν υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Το M. Τζούρι 18, 17, 19 δεν θα ψηφιστούν. Η 124 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 125-126 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός ο, μικρόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 139 υπέρ κατά αποχές Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Απορρίφθηκε πράγματι. Λοιπόν, η 142 υπέρ. 142 κατά. Είναι πολύ δύσκολο να δει κανεί τι γίνεται αν δεν συμμετέχουν τα μέλη του ΕΛΚΑ. 142 και πάλι υπέρ κατά αποχές δεκτή οι υπόλοιπες καταπίπτουν και περνάμε στην 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τζουρί 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τζουρί 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ε, εντάξει, ναι. Διαδικαστικό. Μια ερώτηση για διευκρίνηση. Στον συμβιβασμό H υπήρχε μια προφορική τροποποίηση που είχε προβλεφθεί στον συμβιβασμό. Υποθέτω ότι ψηφίστηκε από κοινού με το συμβιβαστικό. Ήθελα να είμαι βέβαιος γι' αυτό. Με διαβεβαιώνετε. Πιθανότατα θα έπρεπε να το, είχα αναφέρει, να το είχα αναφέρει. Μάλιστα είναι εδώ. Κανένας δεν είχε κάποια αντίρρηση. Δεν είναι γι' αυτό. Εντάξει λοιπόν. Ψηφίζουμε τώρα το τελικό κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Μάλιστα. Oh. Πώς καταφέραμε αυτό να ακυρωθεί. Μα ψηφίσαμε την αιτιολογική σκέψη 1. Α, δεν, το ψηφίσαμε στο αρχικό κείμενο. Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Σκεπτικό 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα τελική ψηφοφορία στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε και πάλι. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Να, ψηφ... να προσθεθούν δύο εντάξει έστω. 38 λοιπόν υπέρ τρεις εναντίον δύο αποχές. Πολύ καλά. Και περνάμε τώρα στη συνέχεια. Στο επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία για το διορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Πίτερ Πράτ. Είχαμε την ακρόαση σήμερα το πρωί. Συμφωνείτε διαβοής να συμφωνήσουμε, ναι. Ωραία, λοιπόν. Ε, διαβοής, να ακούσω. <laughs> right, that's done. Καλώς. Συμφωνήσαμε λοιπόν, εγκρίθηκε. Και περνάμε στο σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κούτας για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ετήσια εκθεσή τη. Τροπολογία 2 υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, Ξανά. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονικά. Πρέπει να ελέγξουμε παρόλα αυτά. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 18 καταπίπτει. Συμβιβαστική γάμα τώρα. Σι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D, δέλτα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 31 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της Απορρίπτεται. Απορρίπτεται παρόλα αυτά. Αρχικό κείμενο, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, δεν είπε ο πρόεδρος, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της 31. Όχι. Είναι το δεύτερο τμήμα του αρχικού κειμένου της παραγράφου 11. Ωραία, ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Άρα είχα δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε ή αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 37 έχει αποσυρθεί. Αρχικό κείμενο τότε της παραγράφου 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F σίγματα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, 39. Ψηφίστε παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 40. Α, όχι, καταπίπτει 40. Το αρχικό κείμενο της 40 τότε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 πίπτη, 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται συμβαστική GZ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ. Παρακαλώ, ο κύριος Ελκατραβή Στο κατάλογο ψηφοφορίας βλέπω ότι για τις 48 και τις 49 είναι συμβατέ ω προστίκη, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε τη 48 και την 49. Α, συμπεριλαμβάνονται στο συμβασμό. Εντάξει τότε. Ναι, ναι, ήταν για την περίπτωση που απορρίπτωταν ο 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ, κατά απόχέ, εγκρίνεται, 52 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται, 52 να ελέγξουμε. Εντάξει, πολλά χέρια δεν σηκώνονται, αλλά εντάξει. Ψηφίστε. Κύριε Θεό, τι ψηφίζετε. Κύριε Κίκολ. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 21. Υπέρ παρακαλώ. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Α, κατά τμήματα. Μάλιστα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά για την τροπολογία 53 παρακαλώ ψηφίστε. Εγκρίνεται. Το πρώτο. Δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γνωμοδότηση κοντ. 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, α... ακαλύπτεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5. Υπέρ, Μέχρι και τη 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 15, κόντ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Και εγκρίνεται. Τώρα δεν τελειώσαμε. Ψηφίζουμε το κείμενο ψηφίσματος. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίζετε παρακαλώ είσαστε διάφοροι εκεί που έχετε τις κάρτες σας στο μηχάνημα χωρίς να πατάτε το κουμπί. Ψηφίστε. Άλλοι έξι μένουν. Πέντε. Πέντε πρέπει να ψηφίσετε ακόμα. Τέσσερις. Τρεις. Δύο. Ένας. Κάποιος δεν θέλει να ψηφίσει. Καλά. Τι να κάνουμε. Πέρα τη ψηφοφορίες. 31 ψήφοι υπέρ. Yes, yes. Voilà. So this is the first vote and then the second. What do you mean? There is a second vote, which is this. Yeah. It's nothing. Okay. okay. Now we go. Συνεχίζουμε τώρα. Και περάμε επαγγελματική διασυνοριακή μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ. Τροπολογία 3. Υπέρ. 3 με 7 unblock μαζί. Εντάξει, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπόλοιπες 8 και η προφορική μαζί, όλες μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. 35, ομόφωνα, μπράβο. Συγχαρητήρια και το, νομοθετικό, το κείμενο νομοθετικού χαρακτήρα, παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίστε. Σας παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ, λέει η πρόεδρος. Πατήστε το κουμπί. Άλλοι τέσσερις μένουν που δεν έχουν ψηφίσει. Δύο. Καλά, κλείνω την ψηφοφορία. 34 υπέρ. Τώρα, Συνεχίζουμε και ψηφίζουμε την έκθεση της κυρίας Σοφία Κονή. Εδώ μία ψηφοφορία όλοι και όλοι, αλλά πρέπει να σας το διαβάσω και λέει ότι αυτός ο κανονισμός του Συμβουλίου για τη δικασία έγκρισης έχει να κάνει με την επέκταση του κανονισμού συναπόφασης όσον αφορά την διασυνοριακή μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών ε, και προς τις χώρες που θα το ευρώ. Οι δύο κανονισμοί θα ψηφιστούν στις 16 Μαρτίου. Οπότε εμεί τώρα ψηφίζουμε την επέκταση ηλεκτρονικά. Μία είναι η ψηφοφορία όλοι και όλοι. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ. Συγχαρητήρια κυρία Οκονή. Έχετε μια ψήφο παραπάνω από την προηγούμενη έκθεση. Και τώρα πάλι της κυρίας Οκόνη πρόκειται για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική α. Εδώ έχουμε από την Άλντε μια προφορική τροποποίηση για την συμβαστική α. Hey, ε, συμφωνείτε? Τη δεχόσαστε την προφορική τροποποίηση. Θέλετε να την ψηφίσουμε την προφορική τροποποίηση. Ψηφίζουμε την, τρο... την προφορική τροποποίηση χωριστά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η προφορική τροποποίηση απορρίπτεται. Συνεπώς ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία τώρα. Αριθμός μάλλον α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά καλύτερα. Θα ελέγξουμε. Αρχική συμβιβαστική τροπολογία A, α. Ψηφίσατε όλοι, πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β, β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, με προφορική τροποποίηση του εισηγητή. Πρώτα. Λοιπόν, δύο ψηφοφορίε έχουμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα για την προφορική τροποποίηση του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι ότι έχουμε μια προφορική τροποποίηση στην προφορική τροποποίηση του εισηγητή που πρέπει επίσης να ψηφίσουμε η οποία θέλει να τροποποιήσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αποχές απορρίπτεται. Εύκολο. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Α, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές Για να βλέπω τα χέρια σας παρακαλώ. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίστε. Για η άλλη να δώσει κανένα σχήμα. Παρέμβαση εκτό μικροφώνου, δεν την ακούσαμε. Okay, four of you haven't voted, three, two. Ωραία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ήταν Τώρα, 10. Αρχικό κείμενο, όχι ούτε και αυτό. Τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14, με προφορική τροποποίηση του εισηγητή. Μάλλον τις εισηγήτρια. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 15 έχει φύγει, η 16 έχει αποσυρθεί, η 17 τώρα. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ,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 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, ψηφίστε. Εξαρτάται βέβαια που κάθεται κανείς. Δεν ε, σας βλέπω καλά όλους. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίες, 26 υπέρ εγκρίνεται. Μετά από αυτή την θα έλεγα έντονη ατμόσφαιρα περνάμε στο 8. Επιλογές πολιτικής για την θέσπιση Ευρωπαϊκού Δικαίου Συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Εισηγητής συντάξη νομοδότησης σε Παπίτικάινεν. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Δεν βρίσκεται, δεν παρευρίσκεται. Η κυρία Πιτικάινεν δεν παρίσταται.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 ΣΥΠΑ θα εξετάσουμε τη δική σας νομοδότηση. Θα δούμε τις τροπολογίες. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμη Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν μπορέσαμε να το εξετάσουμε αμέσως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους όμως για την πολύ επικοδομητική συνεργασία και στη συνεργασία και για τις τροπολογίες. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να καταλήξουμε σε ένα πακέτο για τις συμβιβαστικές για τις τροπολογίες που θα τύχανε της ε, έγκρισης ε, της Επιτροπής. Δεν έχουμε κάποια μεγάλα προβλήματα ή θέματα εδώ. Είχαμε σχόλια που εξετάστηκαν για την οδηγία περιπηρεσιών. Κάποιοι συνάδελφοι σε σχέση με αυτήν την αναφορά είχαν διαφορετικές απόψεις και έχουμε και τη γραμμή κατά του να συμπεριληφθούν οι ελληνικές υπηρεσίες στο συμβατικό αυτό δίκαιο, στην πρόταση. Προτού τώρα ε, ακουστούν περαιτέρω σχόλια, θα ήθελα να συνοψίσω τα κυριότερα θέματα για την έκθεση, αν υπάρχει χρόνος. Πρώτον, το συμβατικό δίκαιο είναι μια καλοδεχούμενη πρόταση και έτσι πρέπει να προχωρήσει και να είναι καλή και για την Ευρώπη και τους καταναλωτές και καλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, πρέπει να, υπάρξουν, να υπάρξει μια μελέτη επιπτώσεων ώστε να υπάρξει νομική βεβαιότητα και αποσαφήνιση κάποιων θεμάτων όσον αφορά τα μέσα της ε, ε, opting in δυνατότητας ε, συμμετοχής και πρέπει να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι οποιασδήποτε προτάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις θα πρέπει πρώτον να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όπως αυτή τη στιγμή στην οδηγία περί δικαιωμάτων καταναλωτών σε σχέση με την οδηγία αυτή για την και την έγκριση αυτών των θεμάτων πριν από την λειτουργία αυτού του εγχειρήματο. Και δεύτερον, αν σε μείζωνα θέματα στα κράτη-μέλη η νομοθεσία υπέρ των καταναλωτών προβλέπει υψηλότερο επίπεδο προστασίας, αυτό έχει προτεραιότητα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβατικό Δίκαιο που θα υφίσταται, θα διασφαλίζεται το ανώτατο όμω επίπεδο προστασία καταναλωτών. Δεύτερο σημείο, θέλουμε να ζητηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με τι business to business contracts, συμβόλαια επιχειρήσεων επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμή ήταν διστακτική να συμπεριλάβει και αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για το σημείο για τι τελικέ υπηρεσίε, όπου η παρατήρηση είναι ότι πρώτον φυσικά θα πρέπει να εξετάζονται σε τομεακό επίπεδο από πλευράς νομοθεσίας. Αν θα υπήρχε όμως ε, κάποια περίπτωση όπου θα έπρεπε να υπάρξει συμπερίληψη, ένταξη αυτών όπως σε κάποια ασφαλιστικά θέματα συμβάσεων ή σε σχέση με πιστώσεις ε, για τους καταναλωτές θα πρέπει να υπάρξει πρώτα μία μελέτη επιπτώσεων και μία ομάδα ε, παϊόντων θα πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σκιώδεις εισηγητές που θα ήθελαν να παρέμουν. Σβέν, θέλετε να πείτε κάτι. Κάθριν, εσείς. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή συνάντηση και συνεργασία που είχαμε. Δεν έχω πρόσθετα σχόλια σε αυτή τη φάση. Okay, Catherine. Εντάξει, Κάθριν, εσείς. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Θα έλεγα, πολλή δουλειά έχει επενδυθεί εδώ και σε σχέση και με τις ε, τροπολογίες και τις προτινόμενες ε, συμβαστικές λύσεις που έχει υποβάλει η συγγήτρια, ιδιαίτερα υποστηρίζεται η μελέτη επιπτώσεων. Αυτό που είχαμε συζητήσει και στη συνέντευξη του Στρασβούργου είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν δει κανείς του λόγου, γιατί πολλοί καταναλωτές δεν επιλέγουν, δεν επιλέγουν διασυνοριακά και 72% αναφέρεται σύμφωνα με μια μελέτη. Και αυτό οφείλεται στις τιμές που ε, ισχύουν. Και μόνο ένα ισχυρό ποσοστό είπαν ότι είναι ε, εντάξει, δεν είναι καλό σε αυτό. Πρέπει να κατανοήσουμε απόλυτα τις επιπτώσεις ε, του, τι κάνουμε. Μελέτη επιπτώσεων έχει, είναι μεγάλη σημασία σε αυτό. Και σε σχέση με την ψηφοφορία που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα να ληφθεί υπόψη αυτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σκιώθηση για την άλλη εγώ. Ουσιαστικά δύο σχόλια θα είχα. Το ένα ήδη καλύφθηκε ότι είναι μια opt-in εθελοντική συμμετοχή ως εναλλακτική λύση. Και επειδή θα επιλέγει κανείς για να μπορέσει να στεφθεί με επιτυχία, πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα εθελούσια συμμετοχής, να προσφέρεται αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας που είναι αναγκαίο. Στην δική μου τροπολογία 17 για το opting in, η λέξη therefore θα πρέπει να υπάρχει στο κείμενο και να διαχωρίζεται με ένα κόμμα και από ό,τι κατανόησα σε σχέση με τις συζητήσεις με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων από πλευρά εισηγητού που είχε αναλάβει επί χρόνια το έργο αυτό δεν στόχευε να καλύπτει χρηματοπιστωτικές ε, ε, υπηρεσίες. Ε, πρόκειται για καταναλωτές και μικρότερα, μικρότερου πλαίσιου συμβάσεις και όχι τόσο περίπλοκα θέματα που θα απαιτούσαν πιθανόν μια διαφορετική κάλυψη ή πρόταση. Και έτσι Τούτων λεχθέντων νομίζω αυτό είναι σωστό και ίσως και γι' αυτό κιόλας κάποια μέλη αυτής της Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι διστακτικά και έχουν επιφυλάξει. Αισθάνονται ότι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα να συμπεριληφθούν χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε σε αυτή την πρόταση. Και γι' αυτό αναφέρω ότι ποτέ δεν ήταν αυτό. Αναφέρεται ότι ποτέ δεν, ήταν, δεν ήταν η πρόθεσή μα. Και έτσι λοιπόν αυτά είναι όλα τα όσα είχα να αναφέρω. Σύρπα θα, θα θέλατε να απαντήσετε, να τοποθετηθείτε, ολοκληρώνοντας. Η κυρία Συγχύτρια, νομίζω καλύπτονται έτσι σαφώς τα περισσότερα θέματα με τις απόψεις που εκφράστηκαν. Μία ερώτηση θα είχα για αυτό το θέμα, για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα έπρεπε να αποκλειστούν απόλυτα, έτσι, να αποκλείονται ή θα ήταν δυνατόν να έχουμε κάποια προσέγγιση ότι ναι, μεν σε αυτή τη φάση θα αποκλειστούν, αλλά μακροπρόθεσμα θα υπάρχει δυνατότητα μετά τη μελέτη επιπτώσεων και μετά την ε, πραγματογνωμοσύνη της ομάδας επαϊόντων να επανεξετάσουμε το θέμα και ίσως να, ενταχθούν. Θα ήθελα την άποψή σας επ' αυτού, Πρόεδρος. Πιστεύω ότι θα ήθελα πολύ περισσότερο να εμπλέκεται αυτή η δική μας ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε σχέση με τις διάφορες υπηρεσίες. Ε, υπάρχουν διάφορα είδη συμβάσεων κτλ. Και δεν νομίζω ότι έχει καν συνταχθεί με όλες αυτές τις λεπτομέρειες υπόψη. Και έτσι δεν βλέπω πώς θα μπορούσε μια μελέτη επιπτώσεων να αντιστρέψει αυτό και μια ας το πω έτσι επιστροφή, επαναφορά του θέματος να ικανοποιήσει τα αιτήματα αυτά. Έτσι λοιπόν σε σχέση με το, την συμπερίληψη που ε, σε σχέση με τον εισηγητή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων αναφέρεται μια δυνατότητα σε σχέση με τα ατυχήματα, αυτοκινητικά ατυχήματα ανάλογα με το ποιος οδηγεί, ποιο αυτοκίνητο, σε ποια χώρα και ανάλογα με το τι εφαρμόζεται από πλευράς νομικών διατάξεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους εσείς ε, οδηγείτε ένα αυτοκίνητο αντεμού σε μια χώρα, το ποιος καλύπτει τα βάρη, τα ασφαλιστικά, είναι, ρυθμίζεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Και αυτό είναι το μόνο το οποίο θα μπορούσε να εξεταστεί. Υπήρχε μια, στο πω έτσι, σύγκρουση αρμοδιοτήτων ε, όταν υπευλήθη αυτή η πρόταση. Και εγώ συμφώνησα ότι μόνο αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Θα ήταν ανόητο αν τώρα λέγαμε ότι θέλουμε το σύνολο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό. Λοιπόν, εντάξει, με αυτή τη διαφοροποίηση θα ψηφίσουμε στις 22 Μαρτίου στην Τζούρι στις 11 Απριλίου και στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο θα περάσουμε στη Σύνοδο του Μαΐου. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο το 9 στην ημερήσια διάταξη. <clears throat> Τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων αναδιατύπωση. Πίτερ Σκίνερο εισηγητής. Πίτερ, έτοιμος είσαστε. Εστέ έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η ασφάλιση, η κάλυψη των καταθέσεων ε, για ασφαλιστικά θέματα στην Ευρώπη είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των αγορών ως ένα μέτρο με μια νέα αναδιατύπωση να υπάρξει η δυνατότητα να καταλήξουμε σε ένα πιο σταθερό σύστημα των ε, δυνατοτήτων ε, ασφάλισης των καταθέσεων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό υπέβαλε μια πρόταση που εγώ συμμερίζομαι σε κάποια τμήματα και την αποδέχομαι. Σε κάποια άλλα τμήματα δεν την δέχομαι όμως. Για να είναι σαφής οι διαφοροποιήσεις θα ήθελα πρώτον στις διαφορές προσέγγισης σημασιολογικά να, επισημάνω, να επιστήσω την προσοχή σας και μετά ακολουθούν εξειδικευμένες επιλεπτομεριών ρυθμίσεις. Η προσέγγιση συνολικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει εδώ ουσιαστικά ένα, μία πρόταση που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. One size fits all. Αυτό μετά από πολλές συζητήσεις με πολλούς εκπροσώπους εκπροσώπων ε, τέτοιων ασφαλιστικών οργανισμών, τραπεζών αλλά και κυβερνήσεων από πολυάριθμα κράτη-μέλη, θα έλεγα ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στα κράτη-μέλη. Μια και η διαφοροποίηση σε σχέση με ήδη καλώς λειτουργούντα συστήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη που υπάρχει όπως ε, είναι ανάγκη να γίνεται. Κατανοώ βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέγει ότι χρειαζόμαστε στην Ευρώπη μια, ε, ένα συνολικό ε, ίσο επίπεδο προστασίας ε, καταναλωτών. Αλλά το one size fits all ισοπεδωτικά δεν είναι πιστικό και δεν το δεχόμαστε. Τι θέλουμε. Πρώτον, θέλουμε την ίδια προστασία των, όσον αφορά τους επενδυτές. Δεύτερον, η ίδια σταθερότητα των ασφαλιστικών συστημάτων στην Ευρώπη. Τρίτον, δεν θέλουμε στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών οργανισμών ιδρυμάτων. Αυτά όμως μπορούν και να υλοποιηθούν όταν και αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές οι απαιτήσεις ρυθμιστούν με ένα ίδιο πλαίσιο απαιτήσεων που θα πρέπει να ισχύει πανευρωπαϊκά. Μεταξύ αυτών με την ρύθμιση και σεβασμό όλων αυτών των διατάξεων και κανονισμών αλλά στο επίπεδο των κρατών μελών και έτσι να έχουμε την μέγιστη ελαστικότητα όσον αφορά τον εξοπλισμό της λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Ε, αυτό τι σημαίνει συγκεκριμένα. Σημαίνει ότι στα κράτη-μέλη μελλοντικά σε ένα ευρύ φάσμα από συστήματα paybox που δεν είναι τίποτα άλλο παρά δυνατότητες καταβολής ποσών ε, αντιστάθμισης ε, σε περίπτωση πτώχευσης μέχρι συστημάτων προστασίας όπως στη Γερμανία, Αυστρία και μελλοντικά στην Ιταλία θα υφίσταται προστασίας. Μικτά συστήματα, Δυστυχώ ο συνάδελφο Σάντσες Πρεσέντο δεν είναι εδώ παρόν, το ιδιαίτερα εκτιμόμενο σύστημα της Ισπανίας που μπορούν να παρεμβαίνουν και στην ατομική περίπτωση διάσωσης τραπεζών αλλά και στην ανάγκη να πληρώνουν τις αντισταθμίσεις ε, και τις αποζημιώσεις. Και αυτό είναι δυνατόν. Αυτή η διαφοροποίηση ε, επί της προσέγγισης ε, και στον τομέα της διάσωσης αλλά και στον τομέα της πρόληψης και στις παρεμβάσεις για την δράση του σε αυτόν τον τομέα είναι κύρια διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, στα επιμέρους σημεία, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η δική μου πρόταση εδώ προβλέπει μια πιο ενισχυμένη δυνατότητα χρήσης των κονδυλίων στο, στο επίπεδο πρόληψης, καθώς επίσης και στο επίπεδο διάσωσης επιχειρήσεων. Όλα αυτά όμως όχι σύμφωνα με μια κατατοδοκούν χρήση του συστήματος αυτού, διότι πάντα πρέπει να είναι σαφές και δεδομένο ότι στην επόμενη φάση διάσωσης θα υπάρχουν επαρκή, ταμεία, ε, επαρκή κονδύλια στα ταμεία αυτά για να υπάρξει ε, παρέμβαση διάσωσης. Αλλά πάντα σύμφωνα με κανόνες που σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ισχύουν και που θα εποπτεύονται στο εθνικό επίπεδο από τις εποπτικές αρχές. Μία ελεγχόμενη δηλαδή διάθεση κονδυλίων από το Ταμείο Εγγυήσεων, εγκυοδοσίας δηλαδή, Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξουν πολλές τέτοιες διασωστικές τέτοιες δράσεις, παρεμβάσεις όπως προβλέπεται και από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ίδια σταθερότητα για τα ε, ε, ε, ταμεία ασφάλισης και ίδια προστασία για τους επενδυτές 100.000 ευρώ, ύψους 100.000 ευρώ. Η ίδια όμως ε, θα έλεγα κάλυψη απαιτεί και την ίδια στοχοθέτηση των ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 1,5% όσον αφορά το, το eligible deposits. Εγώ προτείνω 1,5% των καλυπτόμενων αυτών ε, δαπανών. Γιατί το κάνω αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στις ε, συνολικές εγγυήσεις μιας χώρας, λέγοντας ότι σε καμιά χώρα δεν είναι δυνατόν συνολικά μια δεδομένη στιγμή να υπάρχει αθρηστική, αθρηστικά υπολογισμός όλων των ε, κονδυλίων. Διότι υπάρχει και η single customer view για τα επιμέρους άτομα που ε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό θα μπορεί να γίνεται στο άμεσο μέλλον. Σε άλλες χώρες δεν θα μπορεί να γίνεται αυτό. Και γι' αυτό να επιλεγεί τώρα ως βάση υπολογισμού μια βάση που παρεκκλίνει σαφώς από εκείνα που ουσιαστικά θα έπρεπε να ληφθεί ως βάση υπολογισμών δεν θα ήταν λογικό για να, ε, ε, να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους επενδυτές. Δεν θα ήταν λογικό γιατί. Διότι αυτό θα οδηγούσε σε τελείως διαφορετική σταθερότητα των διαφορετικών πυλώνων ασφάλισης. Όταν βλέπουμε τα αριθμητικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το 1,5% όσον αφορά τις ε, ε, εγγύσιμες ε, δαπάνες έναντι όλων των δαπανών που προτείνω εγώ με 1,5% θα καταλήγαμε σε 23% στην Ολλανδία για παράδειγμα. Δηλαδή θα πληρώνουν πολύ περισσότερο στο Λουξεμβούργο για την σταθερότητα και αν θέλουμε να έχουμε μια παρόμοια σταθερότητα των πυλώνων στην Ευρώπη πρέπει οι εγγυήσει για την κάλυψη αυτών των κινδύνων να υπολογίζουν και να προέρχονται από το Ταμείο Ασφαλίσεων. Και αυτό δεν είναι τίποτα μαγικό. Το απέδειξε το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι θέμα σωστών υπολογισμών και στελεχών. Και γιατί δεν το κάνουν αυτά, αυτό τα ε, ιδρύματα Εγγύσεων Λένε ότι αυτό όταν εμείς πτωχεύσουμε δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει περαιτέρω. Εγώ όμω σε αυτό το σημείο, στην έκθεσή μου, επιλέγω μία προσέγγιση που θα είναι κίνητρο. Κίνητρο ακριβώς για την μετατροπή των καλυπτόμενων αυτών εγγύσεων το δυνατόν νωρίτερα κιόλα χρονικά. Και γι' αυτό προτείνω, γνωρίζοντα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσφέρουμε την κάλυψη αυτή, λέμε ότι από πλευρά αρχή 1,5% των καλυπτόμενων εγγύσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Συστήματα που δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό θα πληρώνουν το ίδιο ποσοστό, αλλά για το σύνολο των eligible deposits έτσι θα είναι πιο ακριβό, πιο δαπανηρό αυτό για συστήματα που δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν τις αναγκαίες ε, εγγυήσεις έτσι θα δημιουργηθεί υψηλό κίνητρο για τις αγορές να πορευθούν προς αυτή την κατεύθυνση των δυνατών γοργότερα, να υιοθετήσουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα covered deposits να μπορούν να προσφερθούν στους επιμέρους καταναλωτές. Γιατί θα είναι αυτό πιο ευνοϊκό για αυτά τα ιδρύματα. Και το Ηνωμένο Βασίλειο απέδειξε ότι μπορεί γοργά να υλοποιηθεί ένας τέτοιος στόχος. Σημαντικός είναι ο στόχος αυτός για τα covered deposits και την single customer view. Ιδιαίτερα όμως και για για το θέμα των διοριών πληρωμών των αποζημιώσεων αν υπάρξουν προβλήματα. Προβλέψαμε μέχρι τώρα 20 20 ημέρες και αν χρειαστεί άλλες 10, δηλαδή σύνολο 30 ημερών ως διορία. 20 ημέρες για την καταβολή του ποσού αυτού. Όλα αυτά πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να είναι λειτουργικά διότι δεν μπορεί να απαιτήσει κανείς να αναμένουν οι καταναλωτές 20 ολόκληρες μέρες μέχρι ότου τους διατεθούν ε, χρήματα και ιδιαίτερα όταν ε, έχουν ένα κοινωνικό, τομή, ε, ένα ε, κοινωνικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι και χωρίς εντάσεις. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες να συντμηθεί αυτή η περίοδος, αυτή η διορία. Το βρίσκω καλό αυτό ο στόχο. Όμως επειδή δεν έχουμε συνολική εποπτεία του τι γίνεται με το Single Customer View και τα Covered Deposits, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν αυτό να λειτουργήσει ούτε και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εξεταστεί αν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό, σαν συνέπεια όλων αυτών, πρέπει να σταθμίσουμε μεταξύ του συμφέροντο του πελάτη να έχει ταχεία καταβολή των ποσών αυτών και μεταξύ της μη παραπλάνησης του πελάτη μέσω υποσχέσεων που θα μπορούσαν να είναι παραπλανητικές. Λοιπόν, αν έχουμε σε μια αμφιβολία, σοβαρή περίπτωση, πρόβλημα τήρησης αυτών των υποσχέσεων, θα είχαμε πελάτες άλλων τομέων που θα αντιμετώπιζαν κρίσεις ως μόνη δυνατότητα να προστρέξουν στην τράπεζα για να σηκώσουν χρήματα, να πάρουν χρήματα από αυτές, διότι θα εξαφανιστεί η εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αν παρόλες τις δεσμεύσεις δεν μπορούν να καταβληθούν αυτά τα ποσά μέσα στην προβλεπόμενη διορία. Πρέπει να βρούμε την ταχύτερη οδό μεταξύ της γοργότερης καταβολής των ποσών και της ε, ε δυνατότητας να ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους αυτά τα ιδρύματα. Προτείνω λοιπόν εγώ το εξή. Θα ενταχθεί μια ε, διορία καταβολής αυτών των ποσών σε 7 ημέρες. Μια εβδομάδα δηλαδή. Συστήματα τα οποία δεν θα είναι σε θέση να πράξουν τούτο θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι τα τέλη του έτους 2016 να υιοθετήσουν να ε, λειτουργήσουν μέσα σε μια διορία 20 ημερών. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εγγυώνται ότι οι πελάτες τους μέσα στα, στις πρώτες πέντε ημέρες θα μπορούν μέχρι ενός ύψους 5.000 ευρώ να ανακτήσουν τα ποσά τους χωρίς περαιτέρω ε, σε λεπτομέρειες εξέταση των περιπτώσεών τους. Δηλαδή γοργά χρήμα το οποίο θα διατίθεται στον ε, ε, καταναλωτή μέσα σε μια διορία 20 ημερών. Έτσι οι επιπλέον εργασίες μπορούν μέσα σε μια διορία 20 ημερών να καλυφθούν χωρίς πρόσθετες δαπάνες. Εδώ όμως θα έλεγα έχουμε και ένα πρόσθετο κίνητρο το οποίο δημιουργείται για συστήματα των κρατών μελών που δεν είναι σε θέση σήμερα τόσο γοργά να καταβάλουν αυτά τα ποσά να μπορέσουν γοργά να μετατρέψουν και να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ώστε γοργότερα να καταβάλουν αυτά τα ποσά διότι θα είναι δυνατόν να αποφύγουν διπλοεπικαλύψεις δαπανών και θα είναι πιο ευνοϊκό το σύστημα συνολικά για αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε εδώ. Προτείνει παραπέρα αυτή η δυνατότητα λειτουργίας να προβλέπεται και μέσα στο πλαίσιο μιας συνεργασίας των συστημάτων εγκυοδοσίας των ασφαλίσεων στην Ευρώπη. Προβλέπεται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις η υποχρέωση των κρατών μελών να καλύπτουν και να δρούν ως εγγυητές ε, για, για λογαριασμό άλλων κρατών μελών ή δικών τους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όταν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να πω ότι μετά από πολλές εκτενείς συζητήσεις και σε κύκλο συναδέλφων εδώ και σε εκπροσώπηση των κρατών μελών αποκόμισα την εντύπωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν όμως καλή ιδέα. Στην Ευρώπη τι έχουμε. Έχουμε πολυάριθμες διαφορετικές ε, τράπεζες, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποδιαφορετικά πλαίσια λειτουργίας και διαφορετικούς κινδύνους. Εδώ οι πελάτες μιας χώρας ε, για την κάλυψή τους ε, μέσω μιας άλλης χώρας ε, το να ζητηθούν ευθύνες θα ήταν η εσφαλμένη προσέγγιση. Όμως μπορεί να υπάρξει μια τέτοια κατάσταση συστήματα εγκυοδοσίας να έχουν κάποιο συμφέρον να υποστηρίξουν άλλους αν το επιθυμούν. Εδώ αναφέρομαι σε σχέση με τις τράπεζες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην δράση σε σχέση με την Ιρλανδία. Παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει στη ζώνη ευρώ και τις δυνατότητες που είχαν να προστρέξουν και να, είναι, να, να συνδράμουν την Ιρλανδία. Θα πρέπει λοιπόν εθελοντικά να είναι ελεύθερη η δυνατότητα για κάποιες χώρες να παρέχουν πιστώσεις ε, ώστε να λειτουργήσουν τα γεωδοτικά συστήματα άλλων χωρών όταν δημιουργούνται προβλήματα σε σχέση με αυτά και όταν θεωρείται ότι αυτό είναι σκόπιμο και μπορεί να γίνει για λογαριασμό τους. Έτσι η ιδέα αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδυναμώνεται από υποχρέωση που επιβάλλεται υποχρεωτικά σε εθελοντικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν επιθυμεί ο εμπλεκόμενος. Και έχουμε έτσι πάλι προαιρετική δυνατότητα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μπορεί να προαχθεί. Αυτό είναι το ουσιοδέστερο της πρότασής μου. Θα έπρεπε να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη διασυνοριακές τέτοιες δυνατότητες εγγύησης καταθέσεων να τις προαγάγουν, διότι μπορεί να είναι προς το κοινό συμφέρον διαφορετικές ε, τραπεζικές αγορές να μπορούν να συγκλίνουν και να λειτουργούν από κοινού ώστε να διατίθενται περισσότερα κονδύλια υπέρ ενός κοινού ταμείου, δηλαδή μεγαλύτερο ποσό για αποζημιώσεις σε περίπτωση πτωχεύσεων. Από την άλλη όμως πλευρά να μπορούν να εξετάζονται και οι δυνατότητες ε, των χρηματοπιστωτικών αγορών που είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν καλά. Αυτά όμως πάντα με εθελοντική βάση λειτουργίας και όχι υποχρεωτικά για τους εμπλεκόμενους. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να από εισαγωγή να ολοκληρώσω την εισαγωγή μου, αλλά να επιστήσω την προσοχή σε ένα πράγμα. Εδώ για μια ρύθμιση που έχουμε για την ε, Νορβηγία ξεχωριστά, βλέποντα αυτήν, αλλά όλοι οι σκιώδει εισηγητέ πρέπει να πω, πρέπει να, ευχαρισ... να... να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει εισηγητέ για την πολύ θετική συνεργασία του, πολύ επικοδομητική συνεργασία του σε αυτό το σημείο. Τακτικά, σε τακτά διαστήματα με του σκιώδει εισηγητέ όλων των κομμάτων, πριν από την σύνταξη της έκθεσής μου ε, είχα ανταλλάξει απόψεις διότι στόχος μου είναι με, ένα τέτοιο, με μια τέτοια αλλαγή υποδείγματος ε, προτύπου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θετικά σε σχέση με τα κράτη-μέλη και είναι θετικό να ληφθούν υπόψη έγκαιρα και οι προτάσεις των συναδέλφων. Ελπίζω με τη δική μου πρόταση στην έκθεσή μου το έκανα αυτό, να το έχω καταφέρει γιατί κατά τα άλλα θα ακούσω τις παρεμβάσεις σας και θα τις λάβω υπόψη συνέχεια. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Οι σκιώδεις, τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω πια να προσθέσω πολλά σε αυτά τα οποία προανέφερε ο εισηγητής πιο πριν. Και υπό το δικό μου πρίσμα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, βρίσκεται στη βάση αυτή τη έκθεση πρέπει να χαιρετήσουμε την πρόταση αυτή. Στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν κυρίω μια πλούστευση και μια ένας εναρμονισμός των υφισταμένων συστημάτων και καλύτερη προστασία των επενδυτών. Για την προστασία καταναλωτών και κατά της απλούστευσης δεν έχει κανείς κάποια ένσταση ή αντίρρηση. Και φυσικά εδώ και για την πανευρωπαϊκή εισαγωγή κοινών προδιαγραφών και προτύπων. Όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί θα έλεγα ότι τώρα με αυτόν τον εναρμονισμό δεν θα υπερβάλλουμε, δεν θα ξεπεράσουμε τα ισκαμένα. Υπάρχουν de facto διαφορές μεταξύ των εθνικών χρηματοπιστωτικών συστημάτων και πρέπει αυτά να, αυτές οι διαφορές να αντανακλώνται όπως πρέπει σωστά. Και δεν θα πρέπει χωρίς ε, να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη να καταργηθούν ε, αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα ουσιοδέστερα στοιχεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η προθεσμία καταβολής των ποσών ε, σε περίπτωση αποζημίωσης όπως πρότεινε ο Πέτερ Σκίνερ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εφικτές αυτές οι προτάσεις συνολικά. Μετά το 1,5% της, της καταβολής του αποζημιώσιμου ποσού Μακροπρόθεσμα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι λειτουργικό και δεν είναι όριμη μια τέτοια πρόταση που να βασίζεται σε αυτό. Ο κίνδυνος, η προσέγγιση για τον κίνδυνο ήταν θεωρητικά καλή. Αλλά υπάρχουν διαφορές εδώ μεταξύ των εμπλεκόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αντανακλώνται επαρκώς αυτές οι διαφορές. Επιπλέον, πέρα από αυτό, το μέσο διευκόλυνσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη Δεδομένων των διαφορών των σημερινών συστημάτων νομίζω δεν είναι λειτουργική μια τέτοια πρόταση. Και ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι το ότι οι προσπάθειες εναρμονισμού συνολικά πάνε πολύ πέρα, πολύ ε, μακριά σε σχέση με την, Ευρωπαϊκή, με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε κάποια ελαστικότητα εδώ. Αναφέρθηκε από τον Πέτρα Σκίνερ πώς προτίθεται να επιλύσει αυτά τα προβλήματα και πρόκειται για μια ισόρροπη προσέγγιση που διασφαλίζει τα συμφέροντα και την προστασία των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά όμω δεν υπερβάλλει όσον αφορά τι υποχρεώσει που επιβάλλονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μια καλή ισορροπία μεταξύ εναρμονισμού και ε, ισόρροπη αναλογία. Και έτσι εδώ οι εθνικέ διαφορέ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιομορφίες που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Και εγώ θα ήθελα ρητά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα ο Πέτερ σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές ευθύς εξ αρχής μας είχε συμπεριλάβει στη συνεργασία αυτή για την έκθεσή του και ήταν ανοιχτός ε, για τις απόψεις μας σε όλα τα σημαντικά σημεία και ε, βρήκαν απήχηση οι παρατηρήσεις μας ε, στα σημεία αυτά. Δεν είναι κάτι το αυτονόητο αυτό. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή το υποστηρίζω απόλυτα και είμαι βέβαιος ότι μέχρι τις τελικές τελευταίες λεπτομέρειες στις διαπραγματεύσεις για τις τροπολογίες που έχουμε θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Peter, a question? Okay, first. πρώτα λοιπόν. Εντάξει. Ευχαριστώ και προσθέτω τα λόγια μου στις ευχαριστίες ε, του προλαλήσαντα. Μόνο κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Μικροφωνισμός. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι σαφές ότι η χρηματοοικονομική κρίση στους ε, μέσους καταναλωτές οδήγησε σε μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα και γι' αυτό είναι τώρα σκόπιμο, πολύ σκόπιμο να καταφέρουμε έγκαιρα να καταλήξουμε στην εγκυοδοσία και προστασία των μικρών αυτών από ε, αποταμιευτών και επενδυτών και να διασφαλίσουμε ότι θα προσφέρουμε μια λύση που πανευρωπαϊκά θα μπορέσει να λειτουργήσει ω θέμα αρχή και θα ανταποκρίνεται σε κοινέ αρχέ και προδιαγραφέ. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που θα αναπτύξουμε για την περίπτωση εκείνη που δεν θέλουμε ποτέ να εμφανιστεί και να συμβεί, δηλαδή κάποια κρίση ή καταστροφή Γι' αυτό είναι νομίζω σκόπιμο να πάρουμε αυτά τα τρία τμήματα που προληπτικά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ώστε η χειρότερη περίπτωση να αποτραπεί ω τελική έκβαση. Είναι μια θετική αυτή η προσέγγιση. Paybox ε, στοιχεία, paybox elements όπως εισάγονται εδώ αυτά με τι προτάσει του εισηγητή. Αυτό στη μία ή άλλη περίπτωση πραγματικά θα βοηθούσε, θα βοηθήσει ώστε η ε, μη ρευστότα η πτώχευση να μπορέσει να αποτραπεί η πτώχευση, η χρεοκοπία. Εδώ όμως πρέπει να δούμε όμως και τις εξής ακραίες περιπτώσεις. Αν συμβεί κάτι τέτοιο που θέλουμε να αποφύγουμε, θα υπάρξει μια περίπτωση που δεν θα μπορεί να αποτραπεί. Και έτσι θα υπάρξει στο μέλλον ίσως κάποια περίπτωση όπου παρόλη την δομή αυτού του ε, συστήματος, οι εκατοντάδες αυτές χιλιάδες ε, δεν θα βρίσκονται στην αρχική φάση στη διάθεσή μας από πλευρά του συστήματος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποια χρόνια προθεσμία ώστε να καταλήξουμε σε μια ε, ισχυρή αξιόπιστη βάση λειτουργίας του συστήματος πανευρωπαϊκά τώρα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ξεχωριστέ ιδιομορφίε που υποχρεώνουν τα ταμιευτήρια στην Γερμανία να εγγυώνται για εκατοντάδε χιλιάδε αυτή την εγγυοδότηση. Και όχι τίποτα παραπάνω, διότι έτσι θα αποφύγουμε ένα στοιχείο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που είχαμε στο παρελθόν, de facto. Και έτσι δεν θα υπάρχει αυτή η στρέβλωση. Και αυτό είναι καλό. Εθελοντικά, εθελούσια να μπορούν να πούν ότι θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ως ίδρυμα μεγαλύτερο ποσό, καλό. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό. Αλλά να είναι σαφές ότι η ιδρυματική αυτή, θα έλεγα, κάλυψη ε, διαφοροποιείται και από τους εγγενείς κινδύνους ε, που χαρακτηρίζουν αυτά τα ιδρύματα. Και εδώ υπάρχουν και οι μεγάλες διαφορές που κατέδειξαν οι κρίσεις. Δηλαδή έχουμε κάποιες ε, ε, τράπεζες σε κρατήδια της ε, Γερμανίας που είναι ευπρόσδεκτοι εταίροι όσον αφορά την εγγυοδότηση. Από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι αν σκληρύνουν τα πράγματα δεν έχουν δυνατότητα να διασωθούν αν συμβεί και κάτι πάει στραβά. Κατά τούτο λοιπόν πιστεύω ότι θα επιμεριστεί το έργο στις κρατικές αρχές εποπτείας, να ελέγξουν εκείνες τι συμβαίνει. Αυτή η ιδρυματική κίνδυνη είναι μέσα στο πλαίσιο μιας ομοιογενούς κοινωνίας ή θα έπρεπε ο ένας ή άλλος εταίρος ε, να αποχωρήσουν από αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε μια πρόταση, θα διατυπώσουμε μια πρόταση χωρίς να κατονομάζουμε επιμέρους χρηματοοικονομικά, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δεν είναι δική μας δουλειά να κατονομάσουμε τέτοια ιδρύματα, ούτε έχουμε λεπτομέρειες στα χέρια μας να κάνουμε μια τέτοια δουλειά. Όμως απλά και μόνο πρέπει να επισημαθεί αυτό. Έχουμε και μια ξεχωριστή κατάσταση σε σχέση με στεγαστικά ταμιευτήρια. Στεγαστικά ταμιευτήρια σε σχέση με τις δαπάνες που προκαλούνται μέσω μια τέτοια πρότασης. Θα γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση. Είναι επαρκής ε, σε σχέση με τα όσα απαιτούνται. Θα θεωρηθούν ε, επαρκή ε, τα μέτρα που προτείνονται. Κατά τα άλλα θα έλεγα ότι ο εισηγητής και οι προλαλήσαντες κατά τα άλλα ουσιαστικά κάλυψαν όλα τα σημεία που θα έπρεπε να αναφέρει κανείς με πληρότητα. Και έτσι η άποψη ότι σε κάμποσα χρόνια θα χρειαστούν κάμποσα χρόνια για να καταλήξουμε σε μια πλήρη ε, δυνατότητα ε, καταβολής αυτών των ποσών 5.000 ευρώ σε 5 λέει ημέρες ε, νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές είναι καλές και μπορούν να λειτουργήσουν. Βρισκόμαστε κοντά στο τέρμα, στην τελευταία ευθεία πριν από το τέρμα. Χρειάζεται λεπτό συντονισμό στι λεπτομέρειε. Αλλά προσεγγίζουμε το, την τερματική γραμμή, θα φτάσουμε στη γραμμή και θα κόψουμε το νήμα. Ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστούμε. Ο Σβέν παρακαλώ. Μάλιστα, εγώ δεν θέλω τώρα να προσθέσω πολλά ή να επαναλάβω κάποια πράγματα. Θα ήθελα μόνο κάποια πράγματα να πω που συμπληρωματικά πρέπει να εξεταστούν σε αυτά που ανέφεραν ο εισηγητή και οι προλαλήσαντε. Υπό το δικό μου πρίσμα δείχνει η χρηματοοικονομική κρίση, αλλά επίσης και οι εξηγήσει που δόθηκαν από κάποια κράτη-μέλη, από τις κυβερνήσεις τους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εγκυοδοσία, δείχνουν όλα αυτά πόσο θα έλεγα πρόχειρη ήταν η προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τις αγορές. Ταυτόχρονα όμως έχουμε όσον αφορά την κάλυψη κινδύνων όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα από πλευράς εγκυοδοσίας έχουμε μια ατυχή σύμπτωση ταυτόχρονης δηλαδή σύμπτωσης και συγκυρίας ότι έχουμε ε, ποσά ε, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εκατό χιλιάδων ή πενήντα χιλιάδων ευρώ μέσω της ε, διασφάλισης των deposit guarantees. Από την άλλη πλευρά όταν έχουμε το θέμα του τι θα γίνει με τις πολύ μεγάλες τράπεζες όπου όλοι γνωρίζουμε ότι αν κάποια από αυτές τις τράπεζες αποτύχει ή χρεοκοπήσει αυτή η αποτυχία θα τεινάξει στον αέρα το χρηματοπιστωτικό σύστημα και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση της αποτυχίας. Σε σχέση δηλαδή με το πλαίσιο του banking resolution, δηλαδή της επίλυσης χρηματοπιστωτικών προβλημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρέπει να αγοράσει κανείς ε, γουρούνι στο σακί, δηλαδή χωρίς να ξέρει τι θα γίνει στη συνέχεια, πώς θα διασφαλιστούν τα συμφέροντα των πελατών έναντι των τραπεζών και πώς η συνολική σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα διασφαλιστεί. Αυτό είναι μια συγκυρία συμπτωματική των, ε, ε, αυτών των κέριων ε, στοιχείων που δημιουργεί προβλήματα. Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε στο επίπεδο της πρόληψης. Να μην είναι αρνητική η θέση των καταναλωτών αυτών που έχουν επενδύσει κεφάλαια και θα έχουν πρόβλημα να αποζημιωθούν στη συνέχεια. Να μην υποστούν κυρώσεις δηλαδή εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται σωστά. Πρέπει να προσφέρουμε κίνητρα ώστε περισσότερα προληπτικά μέτρα να υιοθετούνται αντί στη συνέχεια να πληρώνουν τα σπασμένα οι αθώοι. Και όσον αφορά την μέχρι σήμερα έκθεση έχω μόνο σε ένα σημαντικό σημείο κάτι να παρατηρήσω και αυτό αφορά το θέμα του αν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ρίζικο spread, η διασπορά κινδύνων είναι επαρκής όσον αφορά τις πραγματικές διαφορές των διαφορετικών κινδύνων, διαφορετικών προτύπων λειτουργίας τραπεζών. Ένα ταμιευτήριο στεγαστικό που έχει διαφορετική ε, λειτουργία, έχει χαμηλότερο, χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου που επομίζεται από μια investment bank, επενδυτική τράπεζα, υψηλού επενδυτικού κινδύνου που δρά και σε αυτόν τον τομέα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πού θα θέσουμε κέντρο βάρους εδώ, στο άρθρο 11 δεν θα πρέπει εκεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση, ότι δηλαδή η διαφορά κινδύνου όσον αφορά τα κεφάλαια κινδύνων θα πρέπει να αντανακλώνται και στο πραγματικό σύστημα ασφάλισης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές και τον ε, εισηγητή τον ίδιο και για τις συζητήσεις που είχαμε για αυτά τα θέματα και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία και πραγματικά δημονώ να ακούσω την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς, πώς προβλέπει την διαμόρφωση αυτού του πλαισίου με τα θέματα του Banking Resolution της επίλυσης των χρηματοπιστωτικών προβλημάτων των τραπεζών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την τεράστια προσπάθεια την οποία έκανε. Υπάρχουν αρκετές διαφορές βέβαια στις, στα προγράμματα εγγυήσεων των καταθέσεων μπορέσαμε να αποφύγουμε στο παρελθόν κάποια σημαντικά προβλήματα και κάποιες συνολικές κρίσεις. Βλέπω ότι δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία ανάμεσα στους, στους κοιόδης εισηγητές εδώ. Το θέμα είναι να δούμε αν θα υπάρξει ε, κάτι το οποίο μας δημιουργεί μια κάποια ανησυχία. Αν υπάρξουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα μέτρα που παίρνει μια χώρα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Είναι κρίμα που δεν έχουμε καταλήξει σαν μια κάποια συμφωνία. Το θέμα είναι παρόλα αυτά και οι υπόλοιπες χώρες να συμφωνήσουν με τις προτάσεις μας. Κάποιοι από εμά πιστεύουν ότι κάποιες από τις προτάσεις ε, όταν χαρακτηρίζονται από γερμανική επιρροή ή από κάποια βρετανική επιρροή θα πρέπει να καταψηφίζονται σώνη και καλά. Εν πάση περιπτώσει για τους χρονισμούς. Πράγματι 20 μέρες είναι πάρα πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. 5 μέρες είναι πολύ μικρή χρονική διάρκεια. Είτε ψηφίσουμε τις 5 και καταλήξουμε στις 7 δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Κατανοώ πλήρως την απόφασή σας ε, να μπορεί κανείς να εισπράξει 5.000 σε μια πάρα πολύ μικρή χρονική περίοδο, αλλά σε επίπεδο πρακτικό. Αυτοί που ελέγχουν ε, τις τράπεζες που υφίστανται πιέσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξουν τους λογαριασμούς, να ελέγξουν ότι ο λογαριασμός δεν είναι αμφισβητούμενος, δεν έχει προηγηθεί σαν παράδειγμα ένα διαζύγιο και δεν χρησιμοποιεί και ο σύζυγός μου ενώ δεν είχε δικαίωμα το ποσό αυτό κτλ. Το 1,5% είναι ένα τεράστιο ε, ποσοστό. Το 1,5% των καταθέσεων. η αδίποτε ανάλυση δεν θα λαμβάνει υπόψη το ότι ήδη ζητάμε από τις τράπεζες να έχουν ένα δίκτυο ασφαλείας και ότι σε σχέση με, το, με την σχέση ανάμεσα στη ρευστότητα και τα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να κατέχουν και την έκθεσή τους να υπάρχει μια σχέση η οποία να είναι εν πάση περιπτώσει δύσκολη για τις τράπεζες και δεν μπορούμε να ζητήσουμε ίσως πολύ περισσότερα. Όπως είπατε βέβαια υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη. Σε κάποιες χώρες μέλη ίσως η χρηματοδότηση να γίνεται εκ των προστέρων και όχι εκ των υστέρων, εξάντε και όχι εξ αλλά αυτό δεν θα ισχύσει και δεν πρέπει να ισχύσει για όλες τις χώρες. Τώρα, για έκτακτες περιπτώσεις, αν κάποιος ε, του καεί το σπίτι, εν περιπτώσει, και πάρει πάρα πολύ μεγάλη αποζημίωση και δεν μπορεί να πάρει τα χρήματά του, προφανώς και θα πρέπει να βοηθηθεί. Και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτούς που έχουν 2 εκατομμύρια λίρες στην τράπεζα να καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο με ένα μικροκαταθέτη. Νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να ζήσει ένα χρόνο και περιμένοντας να υπάρξει ρύθμιση στους λογαριασμούς της τράπεζας που έχει πλέον που είναι σε αδυναμία να δώσει χρήματα. Τώρα, οι διασυνοριακές πληρωμές νομίζω είναι κάτι το οποίο έχει νόημα, θα πρέπει να εξεταστεί. Χαίρομαι που θέσατε το θέμα της Νορβηγίας, ίσως πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι με τους Νορβηγούς είναι λίγες οι τράπεζες ε, που έχουν οι Νορβηγοί, ας τους συμπαθήσουμε λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι εφαρμόζουν τους περισσότερους από τους κανόνες μας και έχουν και υψηλές καταθέσεις. Εφόσον λοιπόν είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και για υψηλές ε, καταθέσεις μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Τώρα για τις τοπικές αρχές. Βλέποντας πώς λειτουργούν ε, τα θέματα αυτά θα θέλαμε οι τοπικοί άρχοντες να φροντίσουν λίγο περισσότερο που βάζουν τα χρήματα. Ε, η δική μου δημοτική αρχή δεν είχε τοποθετήσει τα χρήματά της στην Ισλανδία ή στην ε, ε, καταθετική εταιρεία Northern Rock η οποία εξέπεσε σε εισαγωγικά. Νομίζω επίσης ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Τώρα υπάρχουν και κάποια επιμέρους προβλήματα για τα ονόματα των επιχειρήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα το λύσουμε. Για το θέμα της Γερμανίας. Κατανοώ πλήρως τα δικά σας προγράμματα εγγυήσεων και θέλετε εσείς να υπάρξει πάντα το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης με τις υπόλοιπες χώρες. Αν θέλετε όμως να έχετε ένα αμοιβαίο τέτοιο σχήμα προστασίας το οποίο να βοηθήσει μια εταιρεία να πάρει το κεφόλαιό της από μια τράπεζα η οποία δεν τα πηγαίνει καλά τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με έναν διαφορετικού τύπου κίνδυνο από τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται κανείς όταν χρησιμοποιεί τις λεγόμενες ε, ε, γέφυρες τράπεζες. Εδώ έρχονται οι τροπολογίες 28 και 29. Αν μπορούν αυτές οι αμοιβέ εγγυήσει να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλίσουν τη ρευστότητα των τραπεζών, αυτό είναι διαφορετικό από το να πεις λέγοντας μάλλον ότι ε, κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης περίοδου θα τις χρησιμοποιήσουμε για την παροχή ρευστότητας. Δεν υπάρχει στάθμιση στο 80 σημείο 8 ρευστότητα, ε, εγγύηση μάλλον για ρευστότητα πλήρης. Αν το σύστημα στη Γερμανία επιτρέπει να δίδονται εγγυήσεις ακόμα και σε πιστοτικά ιδρύματα τα οποία δεν αποδίδουν, αυτό σημαίνει ότι θα δεσμεύονται υψηλά κεφάλαια. Και νομίζω ότι οι άλλες χώρες δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα ίσως και να μην σας κατάλαβα πάρα πολύ καλά, προσπάθησα πάντως. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έκανες, ε, Σάιμον. Ένα τελευταίο θέμα, το να είναι όλες οι χώρες ε, μαζί είναι κάτι το θετικό, αλλά είναι κρίμα που η μετάφραση του εγγράφου σου ήρθε σήμερα το πρωί στις άλλες γλώσσες. Πήραμε την Παρασκευή το βράδυ τα αγγλικά, και νομίζω ότι όλο μαζί μας φαίνεται πάρα πολύ γερμανικό σαν απόπειρα. Πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά χρειαζόμαστε όλοι να έχουμε τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή μας. Βέβαια τα γερμανικά μου καλά είναι, κάτι κατάλαβα. Right, have we finished that little... Λοιπόν, τελειώσαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ. Α, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω ότι έχω τον κατάλογο των ομιλητών. Δεν τον αγνοώ, τον σέβομαι. Τα καταφέρνω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ένα σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και υπήρχε στην αρχική οδηγία, είναι το 12.1. 12.1β μικρό. σχετικά με, τις, με τους λογαριασμούς ειδικών περιπτώσεων ή ειδικών συνθήκων και καλύπτεται με τις τροπολογίες 12 και 41. Εδώ έχω μια διαφορετική άποψη από την Βίκη. Επιμένω στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θυμαίνει το πως την προηγούμενη Δευτέρα καθυστερούσαμε και χάσαμε τα αεροπλάνα μας τα μεσάνυχτα γιατί προσπαθούσαμε να το βάλουμε αυτό στα πλαίσια της συνδιαλλαγής. Νομίζω ότι ο περιορισμός σε 12 μήνο μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με κάτι που ονομάζεται λογαριασμός executor, και είναι πάρα πολύ δύσκολο μερικές φορές σε ορισμένες χώρες να καταφέρει κανείς να χρησιμοποιήσει με ταχύτητα ένα τέτοιο λογαριασμό. Οι 12 μήνες λοιπόν είναι ένα θέμα και σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις το θέμα αυτό είναι σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος μπορεί να διαχειρίζεται το λογαριασμό του και να τον μετακινεί, τότε μπορεί να, να ανοίξει 200 λογαριασμούς και να βάλει τα χρήματά του εφόσον έχει πολλά. Αλλά αυτή δεν είναι μία επιλογή για κάποιες περιπτώσεις. Start buying CDSs on a bank. Uh, that's all I've got to say. Δεν έχω κάτι άλλο να πω εδώ. Ο Πίτερ. Δεν θα κάνω αστεία σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Θα είμαι ε, σύντομος. Μετά το Northern Rocks, το Ηνωμένο Βασίλειο Πίτερ, δημιουργήθηκε η εικόνα ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε τράπεζες τις οποίες θεωρούσαμε ότι ήταν αθάνατες παρότι ήταν μικρές βέβαια αλλά θεωρούσαμε ότι ήταν ισχυρές και ε, μπορεί να ήταν μικρές αλλά συλλογικά είχαν πάρα πολύ χρήμα οι τράπεζες αυτές και το ίδιο ισχύει και για τα ταχυδρομεία, για τα ταμιευτήρια μάλλον στην ε, υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς θα τα δούμε αυτά. Μήπως θα μπορέσουμε να σκεφτούμε ότι όλα αυτά απαιτείται να αντιμετωπιστούν με εναρμονισμένο τρόπο σχετικά με την προχρηματοδότηση, το λεγόμενο εξάντεμ, έτσι ώστε οι εγγυήσει ναι με να μην δείχνουν όλες το ίδιο, αλλά να έχουν κάποιες ομοιότητες. Λοιπόν, η ρευστότητα για τέτοιου είδους πιστώσεις που θα προταθούν από κράτες μέλη ε, μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική ε, εικόνα σε κάθε χώρα. Έβλεπα στο Σπίγκελ σήμερα λέγοντας ότι η επόμενη ε, δημοσιονομική, η επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα ταμιευτήρια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ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 Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους οι κίνδυνοι δεν καλύπτονται, αλλά δεν είναι και μεγάλοι κίνδυνοι. Θα καταθέσω τροπολογίες για αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη.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 δεν θα πρέπει λοιπόν για να, να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του, ε, του επίπεδου του στόχου τον οποίο θα έχουμε. Σχετικά με τα ποσά τα οποία θα πρέπει να πληρώνονται θα ήθελα να κάνω μια ποσοτική πρόταση. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση εδώ στο 11.3. Δεν μπορώ να του σχολείου, να πω ως σχόλιο αγαπητοί συνάδελφοι κάθε φορά, κάθε φορά όταν κοιτάζω τις βασικές προτάσεις ή κάθε φορά όταν έχουμε προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκομίζω την εντύπωση ότι εργαζόμαστε ενεργά για εκείνους που δεν, είχαν, δεν έθεταν πρόβλημα μέχρι σήμερα και που καθόλου δεν ασχολούμαστε με εκείνους που αντιμετωπίζουν το κυριότερο ή είναι το κυριότερο πρόβλημα. Και δεν κουράζομαι να απαιτώ όλα όσα κάνουμε για τη ρύθμιση των αγορών αυτών πρέπει να στοχεύουν σε ένα πραγματικό στόχο. Η πραγματική οικονομία να ωφεληθεί, να έχουμε διευκόλυνση πιστώσεων. Οι καταναλωτές να έχουν μια πιο εύκολα ελέγξιμη διαδικασία διάθεσης πιστώσεων και να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για όλα αυτά. Αν γίνεται εδώ μια δημιουργική προσπάθεια που αποτολμούμε, την πολυμορφία του τραπεζικού μας συστήματος προσπαθώντας να την διασφαλίσουμε επειδή αυτή η πολυμορφία και ο πολυσχηδής χαρακτήρας είναι μια ευκαιρία για μας. Γιατί όσο πιο μονολυθικό είναι το πλαίσιο της ρύθμισης των τραπεζικών ιδρυμάτων, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Αν διασφαλίζουμε αυτόν τον πολυσχηδή χαρακτήρα, όμως ταυτόχρονα διασφαλίσουμε τα επίπεδα ασφάλειας ως προδιαγραφές, αυτό θα είναι μεγάλη πρόοδος. Και θέλω να εκφράσω μεγάλο έπαινο προς τον εισηγητή για τις συζητήσεις που είχαμε, γιατί κατάφερε να βρεθεί σε θέση με καινοτόμα προσέγγιση διαφορετικές πτυχές να τις συγχωνεύσει τη μία με την άλλη, ώστε στο τέλος τέλος να έχουμε υψηλότερο επίπεδο προστασίας, μεγαλύτερη λειτουργικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και έτσι αυτή η Επιτροπή μέσω της έκθεσης Πέτερ Σίμων μπορεί να γράψει ιστορία. Πώς με μη αντιπαράθεση, με μη συγκρουσιακό τρόπο μπορούν τα πράγματα αυτά να προχωρήσουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα χαιρόμουν αν είχαμε τη δύναμη να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση και να καταλήξουμε στον στόχο. Αν χρειάζεται ρύθμιση σε κάποιες λεπτομέρειες, όπως χρειάζεται σε κάθε έκθεση, είμαι βέβαιος ότι από κοινού θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό συντονιστής ήδη σήμερα εκφράζω ευχαριστίες στον Πέτερ Ζήμων και για εκείνους που εργάστηκαν δημιουργικά μαζί του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρεται ότι ίσως να θέλουμε να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να, για να υπάρχει συμμεταχείριση των συνομοθετών. Πολύ θα ήθελα να ακούσω πράγματι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει για τα έγγραφα τα οποία έχουν πάει στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Ποιες ιδέες συμπεριλαμβάνονται εκεί. Θα ήθελα επίσης να με επιβεβαιώσετε ότι θα προθεθούν στους δύο συνομοθέτες και θα μας ενημερώσετε για ό,τι με κινήσεις γίνουν. Μπορεί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες για τα έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Έχουν σταλεί φωτοτυπίες στον εισηγητή, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα έχει. Θέλω όμως να αναφερθώ στο ζήτημα που θίξατε, δηλαδή ποια είναι η σχέση ανάμεσα ε, στις ε, τράπεζες και στο σύστημα εγγύσεων καταθέσεων. Υπάρχει ήδη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η πρόταση της Επιτροπής λέει ότι όλα τα ποσά του συστήματος εγγύσεων καταθέσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση της μεταφοράς εγγύσεων προς ένα άλλο πιστοτικό οργανισμό. Ο μόνος περιορισμός από αυτού είναι το payout, η υπόθεση του payout αν μπορούν από άλλες πηγές να έρθουν τα χρήματα ή χρηματοδοτείται καλύτερα πάνω από τον στόχο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η χρηματοδότηση λοιπόν της μεταφοράς είναι ένα τέτοιο μέσο, γιατί τι σημαίνει, σημαίνει ότι οι εγγύσεις καταθέσεων, οι καταθέσεις μάλλον, περνάνε από έναν οργανισμό σε έναν άλλον. Αν υπάρχει συγχώνευση δύο τραπεζών, είτε σε μία από τις δύο, είτε σε τρίτη τράπεζα, τότε ο πιστωτής αλλάζει. Άρα υπάρχει μια μεταφορά των καταθέσεων. Και αν χωριστεί σε, η τράπεζα σε μια καλή και σε μια κακή, η καλή συνεχίζει να εξυπηρετεί τους πελάτες της και μεταφέρεται από μια νομική εντότητα σε μια διαφορετική η κατάθεση. Πάντα έχουμε δηλαδή μεταφορά των καταθέσεων. Αν τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει γίνει μετά την κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται αγορά, οι καταθέσεις βγαίνουν από μία τράπεζα και πάνε σε μια άλλη τράπεζα. Και πάλι έχουμε το ίδιο. Έχουμε μεταφορά των καταθέσεων από μία νομική οντότητα σε μία άλλη. Όλα αυτά καλύπτονται ήδη από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει επικρίσεις και το έχουμε ακούσει και από τις χώρες μέλη και από τους μετόχους ότι δεν ήταν δυνατόν να εγκριθεί η σχετική πρόταση. Είναι προφανές ότι έχουμε για 15 χρόνια τέτοια συστήματα εγγύσεων καταθέσεων. Όμως το Bank Resolution είναι κάτι το οποίο συζητιέται τα τελευταία 2-3 χρόνια μόνο στην Ευρώπη. Συνεπώς χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία, χρειαζόμαστε νούμερα, πρέπει να συμβουλευτούμε τους ε, μετόχους ε, επίσης, αλλά ήταν πράγματα τα οποία τα έχουμε, έχουμε τη σχετική οδηγία ήδη για αρκετό καιρό. Αν οι μέτοχοι, το Κοινοβούλιο ή τα κράτη-μέλη θέλουν να συμμετάσχουν στις δυνάμεις του συστήματος Εκείσων ε, καταθέσεων και του resolution, τότε υπάρχει ήδη στην πρόταση και ευχαρίστως να βοηθήσουμε και εμείς η συνεργασία αυτή να επεκταθεί ώστε η πρόταση για το σύστημα Εκείσων καταθέσεων να μην βρεθεί σε διέξοδο επειδή ορισμένοι λένε δεν θέλουμε τώρα να αποφασίσουμε επειδή ίσως αργότερα να υπάρξουν περισσότερες προϋποθέσεις για το Bank Resolution, για την εξυγίανση τραπεζών. Ευχαρίστως να συνεργαστούμε με τους ε, συνομοθέτες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι τυπικά μπορώ να σας ζητήσω τέτοια έγγραφα στο μέλλον να τα υποβάλλετε πάντα στη γραμματεία της Επιτροπής μας ώστε να είναι βέβαιο ότι θα κυκλοφορήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, του ευρωβουλευτέ. Γιατί όπω θα ακούσατε, υπάρχουν ορισμένοι που δεν είναι εισηγητέ ή δεν είναι σκιώδει και όμω θέλουν να ενημερωθούν και εκείνοι και τα θέλουν τα έγγραφα. Πίτερ, μη μακρηγορήσει, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε άλλα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ολοκληρώνοντα, ευχαριστώ θερμά για τι παρεμβάσει εδώ και που όπως διατυπώθηκαν. Κάποια σύντομα σχόλια για τα επιμέρους σημεία που αναφέρθηκαν. Το γεγονός ότι εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια υποψία σε σχέση με τις γερμανοβρετανικές προσπάθειες. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ε, και μια μικρή επίκριση για τη συμπερίληψη δήμων και κοινοτήτων σε αυτή την προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο προστασίας ε, του νόμου και από τη Γαλλία μπορεί να το δει κανείς αυτό όπου κοινότητες με 50 κατοίκους ε, έχουν διαφορετική α το πω έτσι αντιμετώπιση. Ξέρουμε ότι στη Γερμανία έχουμε μικρές μονάδες που όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν μια καλύτερη προστασία όπως ε, κάθε ε, ε, επενδυτής. Τώρα, όσον αφορά το ύψος της τελικής κάλυψης, αναφέρθηκε 1,5% θα μπορούσαμε σε σχέση με το συνολικό ποσό να πούμε ότι αυτό είναι υπερβολικά υψηλή η ρύθμιση. Η πρότασή μου προβλέπει για 15 χρόνια να επιτύχουμε το 1,5%. Συζητείτε στο Συμβούλιο 1,0% να ληφθεί υπόψη ως ποσοστό για τη συνολική εγγύηση, ώστε η επιβάρυνση των τραπεζών να είναι μικρότερη. Το κατανοώ ότι θέλουμε να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ότι δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε υπερβολική επιβάρυνση για να αποφευθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά μικρότερα αδύναμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να υπάρξει μικρότερη επιβάρυνση ώστε να ληφθεί υπόψη η διαφορά έναντι των μεγαλύτερων ε, ιδρυμάτων. Πρέπει να αποφύγουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Όμως έναντι των μεγάλων τραπεζών πρέπει στον ευρωπαϊκό χώρο να υπάρξει μια ε, ρύθμιση που θα λαμβάνει υπόψη το μέγεθο τους. Να λάβουμε όμω υπόψη ότι ο στόχο μα ε, είναι να διασφαλίζουμε την καλύτερη κάλυψη, όχι την τέλεια, αλλά την καλύτερη δυνατή σταθερότητα σε σχέση με την εγκυοδοσία των καταθέσεων που τώρα θεσπίζουμε ως σύστημα και αυτή η βέλτιστη σταθερότητα, σταθεροποίηση απαιτεί διάθεση κονδυλίων. Και τώρα αν πούμε να μην δεχτούμε το 1,5 και να καταλήξουμε στο 1,0% τότε το ταμείο θα γίνει κατά 1 τρίτο μικρότερο, θα συρρυκνωθεί κατά 1 τρίτο. Νομίζω μια βιώσιμη πορεία είναι αυτή που πρότεινα εγώ. Σε 15 χρόνια να ε, ε, έχουμε την ε, διαμόρφωση αυτού του ταμείου και όχι σε 10 χρόνια. Αυτό τη γραμμική ας το πω έτσι ανάπτυξη του ταμείου την επιτρέπει μέχρι να φτάσουμε στο 1,5%. 15 χρόνια. Κάθε χρόνο θα μεγαλώνει το ποσό ώστε να καταλήξουμε στο τέλος στο 1,0% στο οποίο ε, κάποιοι ήθελαν να καταλήξουν. Θα έχουμε ε, μεγαλύτερη διάρκεια συσσόρευσης ποσών ε, με την μικρότερη, ας το πω έτσι, χρηματοδότηση του 1% αλλά θα καταλήγαμε στο 1,5% και να βρούμε το, την δυνατότητα να είναι βιώσιμο το σύστημα. Μας έδειξε ένα πράγμα αυτή η κρίση στο τέλος τέλος. Ακούστηκαν κάποια καλά λόγια που μπορούν ίσως να καθησυχάσουν κάποιους. Όμως θα έλεγα η ασφάλεια ασφάλεια τελικά για το χρήμα, ότι θα είναι διαθέσιμο το χρήμα αυτό, ακόμα και αν καταλήγαμε σε μια μεγαλύτερη κρίση, πρέπει να προετοιμάσουμε, να προλιάνουμε το έδαφος και να δούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες σήμερα, ώστε σε μια περίοδο κρίσης δεν θα μπορούσαν κάποιοι να ανταποκριθούν και να καλύψουν τις ε, απαιτήσει. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, διότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα ήταν σε θέση να πληρώσουν, ενώ θα είχαν τη βούληση να πληρώσουν. Πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς θα υπάρξει, θα υπάρξει αποταμίευση. Κάθε πολίτης, κάθε άτομο προσπαθεί να αποταμιεύσει, συνάπτει συμβόλαια, προσπαθεί να προχωρήσει έτσι. Οι τράπεζες θα έπρεπε με τον ίδιο λογικό τρόπο, με τον κοινό νου να δράσουν όπως και οι πολίτες, προσπαθώντας να αποταμιεύσουν και εκείνες τέτοιου είδους κονδύλια. Δύο τελευταία λόγια σύντομα για το θέμα του υπολογισμού της συνεισφοράς των επιμέρους τραπεζών. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια πρόταση που εγώ την αποδέχομαι. Όμως μόνο την δέχομαι σε μεγάλο βαθμό αλλά ως πρότυπο που μπορεί να υιοθετηθεί, που μπορεί να υιοθετηθεί από μια χώρα για να υπολογίζεται ποια ποσά μέσα στο πλαίσιο του 1,5% από κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να συνεισφέρονται. Ποια ποσά θα συνεισφέρονται ώστε να γεμίσει το, ταμείο, ο κορβανάς. Πιστεύω ότι οι αγορές οι τραπεζικές στην Ευρώπη είναι τόσο διαφορετικές ώστε και εδώ πρέπει να αφήσουμε μεγαλύτερο περιθώριο για την ελαστικότητα. Ε, ε, γνώρισα κάποιες ε, ε περιπτώσεις τραπεζών τους τελευταίους 7 μήνες που θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω βαρετές που έχουν ένα ε, ε, επίπεδο κινδύνου που δεν αφήνει περιθώρια προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν όμως με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσει κανείς και δούμε τα trade unions από τη μια μεριά και από την άλλη πλευρά την Royal Bank of Scotland τότε διαρωτώ με η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο spread αυτό στο εύρος ταιριάζει για τις διαφορετικές αυτές ανάγκες και καταστάσεις. Γι' αυτό στην παράγραφο 11 στο εδάφιο 3 προβλέπουμε την δυνατότητα για τα κράτη-μέλη εδώ να έχουν μεγαλύτερο spread, μεγαλύτερο εύρος δράσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο κινδύνου για τα κεφάλαια των τραπεζών τους από 10 έως 300 ή από 10 έως 350. Είναι κάτι που πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη-μέλη. Αυτό όμως είναι αυθαίρετο, έτσι δεν είναι. Ανταποκρίνεται όμως στις απαιτήσει και ανάγκες του εδαφίου 11, όπως προ του, παραγρα... άρθρου 11 του αντίστοιχου εδαφίου, με ποια βάση θα πρέπει οι συνεισφορέ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με ένα τέτοιο πρότυπο που θα υιοθετηθεί. Έτσι, με μια σταθερή τροχιά, σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θα μπορούμε να λειτουργήσουμε, αλλά και πάλι με τη μέγιστη δυνατή ελαστικότητα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 31 Μαρτίου. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 20 Απριλίου. Ε, στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Σημείο 17 τώρα στην ημερήσια διάταξη που είναι τα συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων. Ο Πίτερ Σκίνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. ερχόμαστε μετά το σύστημα εγγύσεων ε, καταθέσεων. Τώρα έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ξέρετε. Βέβαια, ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιο σύστημα εγγύησης ασφαλίσεων. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, στο σημερινό οικονομικό κόσμο, ο κόσμος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια κάποια εγγύηση ασφαλίσεων Αυτό σημαίνει για ορισμένου ότι πρόκειται για τις αποταμιεύσει μια ζωής που βάζουν στι ασφαλίσεις. Μπορεί να δει κανεί τι έγινε και με την Equitable Life, που είναι μια πρόσφατη εμπειρία που έχουμε στην πολιτική μα ζωή, όπου οι καταθέτες σε κάποιε χώρες ε, μέλη δυσκολεύτηκαν να βρουν ότι ποιο τελικά ευθύνεται, ποιο είναι ο ρυθμιστής και πού να πάνε να ζητήσουν τα λεφτά του. Έχουμε προνομιούχο ρόλο εδώ Προσπαθούμε να βάλουμε κάποια τάξη σε αυτό το τομέα. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει σε πολλά σημεία προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά τα σημεία. Έχω όμως και κάποιες διαφορές. Είναι σωστό να έχουμε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το στάδιο αλλά να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύσεων ασφαλίσεων. Όπως ακούσαμε και από τον προηγούμενο εισηγητή, είπε ότι οι διαφορές που υπάρχουν οδηγούν σε κάποια αποτυχία. Και είναι δύσκολο να καλυφθούν αυτές οι διαφορές. Καλύτερο όμως σας έχουμε κάτι συντονισμένο, παγιωμένο και σε ένα κάποιο βαθμό να υπάρχουν κοινέ προσδοκίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες μέλη δηλαδή. Πιστεύω επίσης ότι θα έπρεπε να πιέσουμε και τους ε, επιθεωρητές στα κράτη-μέλη. Μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κάθε επιθεωρητής στις χώρες μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνο και πρέπει να μπορεί να ελέγξει τι γίνεται κάθε φορά με τις διάφορες ε, εταιρείες, τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό έχει βγει πάντως από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει ε, στα κράτη-μέλη βάσει της οδηγίας Φερεγκιότητα 2. Πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός αναρμόνισης των κανόνων που ισχύουν ώστε αυτά τα εθνικά συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων να είναι καλά δομημένα και να υπάρχει συνοχή βάσει των εμπειριών που έχουμε μέχρι τώρα. Στη Σλοβακία δηλαδή ένας ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει την ίδια εμπειρία. Αν ισχυρίζεται, μάλλον αν ζητάει χρήματα από κάποια τράπεζα κάπου αλλού, από κάποια ασφαλιστική εταιρεία κάπου αλλού η οποία έχει πτωχεύσει, να υπάρχει συνοχή και να υπάρχει και συνοχή και όσον αφορά τα επίπεδα ε, κάλυψης και εγγύσης. 100% βέβαια θα έπρεπε να ήταν ο στόχος, δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ποια, ποιες ασφαλιστικές ε, εταιρείε πάνε καλά, ποιες όχι, αυτά θα πρέπει να τα ξέρει ο ελεγκτής για να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών ε, σε περίπτωση πτώχευσης ασφαλιστικής εταιρείας. Πολλές πτωχεύουν. Θα πρέπει όμως να μπορούν ακόμα να πληρώσουν το κόσμο. Τα πράγματα δεν είναι ίδια όπως είναι και με την τράπεζα που ε, οι τράπεζε θα πρέπει την επόμενη μέρα να βρουν ρευστό και δεν μπορούν. Ενώ με τι ασφαλιστικέ εταιρείε θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί μπορούν να διαπραγματευτούν και να ανταποκριθούν στι υποχρώσει του απέναντι στου πελάτε του πρέπει να βρούνε βέβαια, κεφάλαιο με κάποιον άλλο τρόπο ασφαλιστικές εταιρείε, εφόσον εννοείται ότι δεν πρόκειται να έχουν νέους ε, πελάτες μετά την πτώχευσή τους. Ξέρετε ότι υπάρχει και το θέμα της αναλογικότητας για το οποίο τσακωνόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάποια όρια. Δεν έχουμε όμως τους ορισμούς που θέλουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξέρουμε πώς επηρεάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε τι αναλογία. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να μπορεί κάποια άλλη στιγμή να μας κάνει καινούργιες προτάσεις. Προς το παρόν πάντως δεν βλέπω πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνώ πάντως για το upfront, εξάντε πόρους που λέει η Επιτροπή. Ποσά τα οποία υπάρχουν για την ασφάλιση και να μπορούν τα χρήματα αυτά να τα πάρουν οι πελάτες τους σε πολλές χώρες δεν ε, αναφέρονται σαν προκαταβολή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν ρεαλιστικό κάτι τέτοιο. Η χρηματοδότηση τώρα των συστημάτων εγγύησης ασφαλίσεων βασίζεται στην επικουρικότητα και ίσως έτσι θα έπρεπε και να παραμείνουν. Αρκεί η εμπειρία του καταναλωτή να είναι ίδια. Δεν έχει σημασία πώς λειτουργεί το σύστημα. Οι κανόνες πρέπει να είναι οι ίδιοι όταν φτάνουμε στον καταναλωτή. Το πνεύμα δηλαδή να είναι το ίδιο. Και το σύστημα εγγύησης να εξυπηρετεί το σκοπό του. Στην έκθεσή μου εγώ μιλάω για τον νέο Ευρωπαϊκό Οργανισμό που θα εξετάζει τα συστήματα και θα κάνει συστάσεις κάθε φορά που τα συστήματα δεν ανταποκρίνονται στο στόχο τους. Θα τονίζουν επίσης τις βέλτιστες πρακτικές, θα ενημερώνουν το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το πώς πρέπει να λειτουργούν. Ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται και τέτοια κεφάλαια για την ε, προχρηματοδότηση των συστημάτων. Βέβαια θέλω τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών και ελπίζω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Jean Paul, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πράγματι. Θα μιλήσω εξ ονόματος του Ότμαρ Κάρας, ο οποίος δουλεύει πολύ αν και είχε προβλήματα μετά το ατύχημά του και μου έστειλε τις σημειώσει του για να κάνω κάποια σχόλια στον Πίτερ. Για τον Ότμαρ Κάρα, στο θέμα της χρηματοδότησης, ο κανονισμός θα πρέπει να σέβεται τα ειδικά χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού τομέα σε κάθε κράτος μέλος και δεν πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. Συμφωνούμε εδώ με τον κύριο Σκίνερ και για την ελάχιστη εναρμόνιση σε σχέση με το ρόλο αυτού του ταμείου, τα συστήματα εγγυήσεων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται παρά σαν τελευταία δυνατότητα. Θα πρέπει να ισχύσει η γεωγραφική ζώνη της χώρας προέλευσης, θα πρέπει να προωθήσουμε τον καταναλωτή και όχι την επιχείρηση και θα πρέπει να περιοριστούμε στις ε, ε, ασφαλίσεις ζωής και όχι στις υπόλοιπες. Ο κύριος Καράς λέει ότι ο κίνδυνος για τον φορολογούμενο θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, η εθνική έλεγχοι και οι κοινοτικοί θα πρέπει να ενισχυθούν, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις αρχές εποπτείας και να εμπλακεί ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλιών και Επαγγελματικών Συνταξιοδοτήσεων. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι μια εξάντε χρηματοδότηση, ο κύριος Κίνερ είναι κατά ο κύριος Καρά θεωρεί πάντω ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να αποφασίζεται στα πλαίσια της επικουρικότητας από τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Καράς ε, εφιστά την προσοχή μας και στα υπόλοιπα θέματα. Η έκθεση Σκίνερ αναφέρεται σε διάφορα μοντέλα και ο κύριος Κάρας θέλει να τα διευκρινίσει είτε με τη δυνατότητα αποζημίωσης του καταναλωτή είτε ε, μέσω της μεταφοράς του συμβολέου σε μια άλλη εταιρεία ασφαλιστική με συνέχιση των εγγυήσεων. Σχετικά με τις λεπτομέρειες και τους ε, ορισμούς κάποια θέματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί σχετικά με τα ε, ενεργά των επιχειρήσεων και τις ευθύνες που προέρχονται από αυτά. Εδώ πάντως δεν χρειάζεται να υπάρξει μια νέα νομοθετική ρύθμιση. Ο κύριος Σκίνερ περιλαμβάνει επίσης και τους ενδιαμέσους ε, του ασφαλιστικού χώρου, αλλά ο κύριος Καράς λέει ότι δεν πρέπει να καλύπτονται από το σύστημα εγγύησεων. Σχετικά με, την, ε, με το όριο ε, για την αποζημίωση, ο κύριος Καράς θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι ειδικέ συνθήκες όταν μια δικαστική διαδικασία σαν παράδειγμα είναι εν εξελίξη και στο τέλος το σύστημα της προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει να εξαιρεί αυτούς οι οποίοι εργάζονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα σχόλια που θέλει να κάνει ο κύριος Καράς και τα οποία σας μετέφερα με προθυμία. Ευχαριστώ. Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και θένα Πίτερ. Όπως πάντα, έκανε μια εξαιρετική δουλειά και εγώ προσπάθησα να βρω κάποια προβλήματα στην έκθεσή σου, στην πρόταση την οποία κάνεις. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία το να αναφέρεις ότι οι ασφαλείες είναι διαφορετικό συστήματα από ότι τα πιστοτικά ιδρύματα και τα συστήματα εγγύησεων των καταθέσεων. Αν συγκρίνει κανείς τις ε, τρεις διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις μεταξύ τους έχουν σημαντικότατες αποκλήσεις. Νομίζω ότι αυτά όπως το κάνεις άλλωστε θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Να ε, διευκρινίσω εδώ εγώ ότι πιστεύω στην αρχή της χώρας προέλευσης ε, στην ελάχιστη αναρμόνιση η οποία μπορεί να προωθήσει, να, να, να, αυξηθεί μάλλον και να φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο αλλά ένα ελάχιστο επίπεδο είναι το αντικείμενο της εγγύησης. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της εμβέλειας της νομοθετικής αυτής ρύθμισης είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να προσπαθήσουμε να πείσουμε ίσως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι καλύπτεται μέσα στην ισχύ αυτή της πρότασης. Έτσι όπως το συζητήσαμε ε, εμείς και εσείς σχεδόν εμπειρογνώμων πείτε, να δούμε ποιες μορφές ασφάλισης καλύπτονται από αυτές τις εγγυήσεις και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα διάφορα είδη των ασφαλίσεων ζωής που χρησιμοποιούνται σαν συνταξιοδοτικά ταμεία. Γιατί ξέρει κανείς πολύ καλά ότι διαφορετικά συστήματα συντάξεων ισχύουν σε βόρειες χώρες που δημιουργήσαν προβλήματα και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και στο μέλλον προβλήματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να το διευκρινίσουμε την εμβέλεια όπως είπα μιλάτε για προστασία 100% σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα πρέπει να με πείσεις σε σχέση με αυτό γιατί αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Είπες ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η κάλυψη και στις λεγόμενες ενδιάμεσες πωλήσει και ακόμα και στις απατηλές ασφαλιστικές δραστηριότητες. Αυτές δεν καλύπτονται από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου εδώ, γιατί αν εξετάσεις τα σχήματα αποζημίωσης των επενδυτών. Εσείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχετε μια ευρία ερμηνεία κάλυψης του επενδυτή καταναλωτή. Αν θελήσετε να εφαρμόσετε την ίδια αντίληψη για το σύνολο της Ευρώπης, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσετε κάποιες εξηγήσει για να πείσετε. Γιατί κάτι τέτοιο δεν οδηγεί μόνο, δεν καλύπτει μόνο την πτώχευση και τις απάτες αλλά και άλλες καταστάσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς. Ε, παράλληλα νομίζω ότι όταν συζητάμε για τέτοιου είδους απαντήσεις προς τον κύριο Μπούλμαν σαν παράδειγμα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς στην Επιτροπή είναι να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Μπορεί κανείς να το πει αυτό αλλά από την άλλη κάποιοι από μας ή κάποια κομμάτια μας αν θέλετε είναι υπεύθυνοι για τις ενεργειές τους και δεν μπορούμε πάντα εμείς να καλύπτουμε τις ανάγκες όλων. Τώρα για τη χρηματοδότηση. Προσπαθώ να δω τι μπορεί να γίνει με τη χρηματοδότηση στα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών. Και ε, αυτά χρηματοδοτούνται εκ των προτέρων. Έχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών. Κάποια άλλα όργανα έχουν και αυτά αμφιβολίες για τα συστήματα και θα πρέπει οι αμφιβολίες αυτές να μας επηρεάσουν και εδώ στις ασφάλειες. Νομίζω ότι αξίζει να έχουμε περισσότερες ανησυχίες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να δώσει κανείς παραδείγματα, αλλά πόσες είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν πέσει έξω ή έχουν κάνει απάτες κατά τη διάρκεια της τελευταίας περίοδου. Άραγε οι ασφαλιστικές εταιρείες δημιούργησαν προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η απάντηση, τουλάχιστον η απάντηση που εγώ πιστεύω είναι ότι δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι σωστό να προχωρήσουμε ε, σε στάδια και οι κατευθύνσεις τις οποίες προτείνεις είναι σωστές τις θεωρώ σωστές. Όμως, καλό θα ήταν να γίνουν κάποιες τροπολογίες για να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτερες. Sven, okay. Vicky, are you... Μετά είναι η σειρά σου, αλλά εξαφανίστηκε κάποια στιγμή γι' αυτό. Μπορώ να περιμένω, λέει ο Σβέν. Δύο μικρά πραγματάκια για το 100% κάλυψη. Αναρωτιέμαι. Όλοι θα το θέλανε, ιδιαίτερα για τις ασφάλειες ζωής, αλλά μήπως πρέπει να πάμε λίγο παρακάτω. Για το πότε γίνονται οι πληρωμές, το χρονοδιάγραμμα. Συνήθως μπορείτε να έχετε μια επιλογή μεταφοράς του πορτφόλιου σε κάποιον άλλον αντί να πάρετε σε ρευστό το ποσό και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και το τρίτο για τις απάτες και εδώ ίσως θα έπρεπε κάτι να βάλουμε χρειάζεται φερεγγιότητα και πρώτα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί Εντάξει, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, προσβλέποντας το να ξαναεργαστώ μαζί σας για αυτό το θέμα, ήδη είχαμε μια γόνιμη συνεργασία για το πακέτο εποπτείας και ε, συνεργαστήκαμε για ένα παράλληλο πρότυπο για το πρότυπο αποζημίωσης. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν αυτά να λειτουργήσουν και εύχομαι στον ε, Ότμαρ Κάρας θερμή καλή ανάρρωση, σιδερένιος. Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσει να ξανάρθει κοντά μας. Είναι κρίμα αυτό το οποίο του συνέβη με αυτή την επίθεση, αυτόν τον τραυματισμό που υπέστη. Πέρα από αυτά έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι έχουμε μια τάση μια τάση να μην παίρνουμε τα προβλήματα στα σοβαρά τα προβλήματα που ακόμα δεν μας έχουν πλήξει, δεν μας έχουν χτυπήσει. Και αυτό είναι μέρος αυτού του προβλήματος σε αυτή τη συζήτηση εδώ. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα και οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρίσκονται γενικά να έχουν το ρόλο των καλών παιδιών. Συμφωνώ, είναι διαφορετικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών από τα τραπεζικά ιδρύματα και σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους. Πρέπει διαφορετικά οι τράπεζες να αντιμετωπίζονται από τα ασφαλιστικά ιδρύματα. Ταυτόχρονα όμως να μην μυθοποιούμε τα πράγματα, μην δημιουργούμε μύθους. Ένας από αυτούς τους μύθους, θεωρώ εγώ υπό το πρίσμα μου, ότι δεν έχει καμιά σχέση με την κρίση, λένε αυτοί, αυτά τα ιδρύματα. Και δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτά τα ιδρύματα λόγω της κρίσης. Να συνειδητοποιήσουμε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή στι αγορέ του ευρώ και να συνειδητοποιήσουμε τι θα γινόταν σε κάποιες ασφαλιστικές αν δεν είχαμε διασώσει τι τράπεζε πιο πριν με τεράστιε παρεμβάσει, χρηματοοικονομικέ παρεμβάσει από πλευρά των κρατών. Τι θα γινόταν με τα ασφαλιστικά αυτά ιδρύματα αν δεν είχαμε διασώσει τι τράπεζε με τεράστιε χρηματοοικονομικέ παρεμβάσει. Καθώ επίση και με πολλέ δημόσιε εγγυήσει. Ακόμα και οι ασφαλιστικέ εταιρείε όσον αφορά τι επενδύσει που είχαν γίνει χωρίς να σκέφτονται πολύ τους ενδυνάμει κινδύνους στις επισφαλείς αγορές θα μπορούσαν να είχαν καταλήξει σε τεράστια προβλήματα αν δεν είχαμε κάνει αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνεται να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή δημόσια κονδύλια για να αντιμετωπιστούν προβλήματα ιδιωτικών τραπεζών σε μια οικονομία της αγοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο συνετοί. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια, θα έλεγα, κάποιος λόγος για τον τραπεζικό τομέα να ληφθεί υπόψη διαφορετικά τα, χρημα... τα ασφαλιστικά ιδρύματα είναι διαφορετικά όμως και πρέπει αυτά να τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και αυτές τις διαφορές. Θα ήθελα σύμφωνα με αυτή την γραμμή τουλάχιστον δύο διαφορετικά θέματα να αναφέρω. Το πρώτο είναι το ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε εγρήγορση όπως και τα άλλα, για τα άλλα δύο συστήματα για τις τράπεζες το όλο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να αποτύχει κάποια μέρα. Δηλαδή για τους εμπλεκόμενους που θα είναι μέρος, μέλος αυτό αυτού του προτύπου ή ήδη είναι μέλη εκεί όπου υπάρχουν τέτοια πρότυπα, τι θα γίνει αν χρεοκοπήσουν ή αν πτώχευαν κάποτε. Και επειδή είναι υπερβολικά μεγάλα αυτά τα ιδρύματα για να τηρήσουν όλα τα υπεσχημένα, όλες τις υποσχέσεις τους θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ καλά και το μέγεθος ως ένα συντελεστή, ως ένα παράγοντα σε αυτά τα πρότυπα που θέλουμε να υιοθετήσουμε. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό να σκεφτεί κανείς για το συνολικό θέμα του ex ante και ex post όσον αφορά την χρηματοδότηση, την κάλυψη των εγγύσεων. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι ότι είναι τόσο σταθερά τα πράγματα στον τομέα των ασφαλίσεων ώστε να πούμε ότι μπορούν να δικαιολογηθούν εκεί απλές εξπόστα post ε, χρηματοδοτήσεις ε, χρηματοοικονομικά και θα έλεγα επίσης υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα κατά αυτής της προσέγγισης. Έχουμε λοιπόν εδώ την περίπτωση μιας ασφαλιστικής εταιρείας που θα πτωχεύσει. Ε, τότε δεν θα συνεισφέρει πλέον με κανένα τρόπο από πλευρά της. Και αυτό είναι με ένα σημαντικό επιχείρημα για μια χρηματοδότηση ex ante, εκ προημίου. Και είναι προκυκλικό επίσης αυτό. Αν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε μια χρηματοοικονομική αγορά και κάνει κανείς τα πάντα ex post, ε, τότε στην περίπτωση που θα χτυπηθεί άγρια η αγορά, θα είχε κανείς τεράστιες δυσκολίες να βρει την χρηματοδότηση ex post και την κάλυψη ex post. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να πάρουν αυτά τα προβλήματα σοβαρά. Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι γιατί για τις τράπεζες και για την investment compensation έχουμε το ex ante ως χρηματοδότηση, ως σύστημα. Υπάρχουν λόγοι για το ex ante σύστημα στην χρηματοδότηση. Έχω προβλήματα στον ασφαλιστικό τομέα να έχουμε ex post post, εξ ορισμού, εξ post χρηματοδότηση. Δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Επίσης βλέπω να υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα κάποιο πρόβλημα στο επίπεδο της συνολικής συζήτησης για την ελάχιστη και μέγιστη εναρμόνιση και ε, Προέλευση, χώρας προέλευση και χώρας υποδοχής αφετέρου. Πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση επί τη αρχής. Αν είμαστε υπέρ εναρμόνιση, τότε τα σήμερα διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη θα, θα, θα έχουν διαφορετική μορφή. Αν όμως ταυτόχρονα είμαστε υπέρ, όπως προτείνει ο εισηγητή, μιας ε, ρύθμισης ε, χώρας υποδοχής, τότε στην ίδια την αγορά θα έχουμε τελείως διαφορετικούς εμπλεκόμενους με τελείως διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανάλογα με τη χώρα προέλευσης σε σχέση με τη χώρα υποδοχής και αυτό θα δημιουργεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό εκεί που δεν θα πρέπει να υπάρχει στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Θα έλεγα αν είμαστε υπέρ του ελάχιστου εναρμονισμού χρειάζεται κάποιο μέρος, κάποιο ποσοστό της υιοθέτησης της αρχής της χώρας υποδοχής. Θα ήθελα περισσότερο να εμβαθύνουμε σε αυτά τα πράγματα, να τα εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος στο μέλλον με τους χειώδεις εισηγητές. Και το τελευταίο μου θέμα θα αναφερόταν στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η Sharon Bowles επεσήμανε πιο πριν. Και ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στην έκθεση ότι καλύπτοντας ε, άτομα, φυσικά άτομα, δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε ως στόχο. Αν υπάρχουν κάποια άλλα επιχειρήματα, Πίτερ, θα ήθελα να μας τα εκθέσεις και ίσως να αναφέρουμε τις αναγκαίες νομικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, ώστε κάτι τέτοιο να καταστεί εφικτό ως θέση. Αυτές είναι οι πρώτες μου αρχικές παρατηρήσεις και αρχικά σχόλια. Αυτό θα, το οποίο θα με ενδιέφερε περισσότερο να συνοψίσω θέλω, είναι να διασφαλίσουμε ότι στο τέλος τέλος η αυτά τα συστήματα βασικά θα είναι εξ άντε στη χρηματοδότηση. Εξ άντε. Σύμφωνα με το επίπεδο κινδύνου των επιμέρου ασφαλιστικών εταιριών, όπω συζητήσαμε πιο πριν και για τι τράπεζε. Και τρίτον, να λαμβάνονται υπόψη οι συστημικοί κίνδυνοι. Οι συστημικοί κίνδυνοι, εκείνοι που είναι πολύ μεγάλη λόγω μεγέθους ως εταιρείε ή επιχειρήσεις να δούμε ότι η ενδυνάμει πτώχευσή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται από δημόσια κονδύλια και αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται με υψηλότερη συνεισφορά από πλευράς τους, χρηματοοικονομική συνεισφορά σε αυτά τα ταμεία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη συνετές αρχές οικονομικής λειτουργίας και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα βρούμε τις σωστές λύσεις. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνεργασία σα. Λυπάμαι που άκουσα ότι είναι αδιάθετος ο κύριος Καράς. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Ίσως ο Ζων Πολ να με ενημερώσει. Πράγματι τα θέματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της ε, μετακίνησης από τη μία εταιρεία στην άλλη των καταναλωτών επενδυτών. Θα τα δούμε αυτά. Σχετικά με την κοινή ευθύνη και γύρω από το αν θα προταθεί ε, θα γίνουν νέες προτάσεις και ε, για να καλυφθούν οι μη ενδιάμεσοι, οι πράκτορες, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Έχουμε κάτι εδώ το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες τις οποίες είχε περιγράψει η οδηγία Solvency 2. ο κύριος Καράς στον συγκεκριμένο τομέα, στον θέμα των ασφαλιών, έχει τεράστια εμπειρία και μπορεί να προβλέψει πάρα πολλά. Τώρα για τα θέματα τα οποία έθεσε ο Σμιτ. Όλοι ευχαριστώ για την υποστήριξή σου, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει τώρα σχετικά με τις απάτες. Ε, υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες, πολλές. Ε, το σώμα είχε περάσει ένα ψήφισμα και νομίζω ότι εγώ δεν πολύ συμφωνούσα, αλλά για μια, ε, ένα ψήφισμα για μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία είχε παραπλανητικές ρυθμίσεις, πουλήσει και συμφωνίες. Ίσως ήταν ανόητοι αυτοί που υπέγραψαν, ίσως ότι δεν πίστευαν ότι μια εταιρεία η οποία έκανε μια υπόσχεση δεν θα την τηρούσε και πίστευαν ότι οι αγορές θα ε, ανέβαιναν συνεχώς, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Λοιπόν, το θέμα των παραπλανητικών πωλήσεων από πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών μακροπρόθεσμα είναι ένα πρόβλημα. Ας προσπαθήσω να το διευκρινίσω κάπως καλύτερα στην πρότασή μου. Θα επανέλθω σύμφωνα πάντο με την περίπτωση της Equitable Life. Θα δούμε αν θα πρέπει να καλύπτονται και εδώ καταθέτες από άλλες χώρες και τα λοιπά, από επενδυτές από άλλες χώρες και τα λοιπά. Υπάρχουν επίσης και αμοιβαίες ασφαλιστικές εταιρείες, υπάρχουν συνεργατικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν καταθέσει τα κεφαλαία τους στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε μια τρομερή ποικιλία η οποία δημιουργεί μια περίπλοκη κατάσταση σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Ξέρουμε ότι οι εταιρείε μέσα στο εσωτερικό μιας χώρας μπορεί να έχουν κάποια ασφαλιστικά κεφάλαια, αλλά μπορεί αυτά τα κεφάλαια να μην τα ε, μεταφέρουν ή να μην μπορούν να τα μεταφέρουν σε άλλες χώρες για εσωτερικούς τους λόγους. Το θέμα είναι να μην ε, επανέλθουμε στις συζητήσεις ε, τις οποίες είχαμε κάνει στα πλαίσια της Solvency 2 όπου προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε μία πρόταση η οποία να στέκει παρά τις διαφορές μας. Εδώ το θέμα μοιάζει με τα πιστοτικά που συζητούσαμε προηγουμένως και τις εγγυήσεις των καταφέσεων. Υπάρχουν πάρα πολλά αντιτιθέμενα συμφέροντα και οι συγκρούσεις θα βγουν στην επιφάνεια. Για τις ευθύνες, πράγματι ε, και εμείς έχουμε ευθύνες, όπως ε, και οι άλλοι εμείς πιστεύουμε ότι για τους πιο ευάλωτους ιδιαίτερα θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας και ε, πράγματι όταν υπάρχει ένα άδικο συμβόλαιο, συμβόλαιο ασφαλιστικό εμείς σαν νομοθέτες θα πρέπει να προσπαθήσουμε τέτοιες καταστάσεις να ε, δημιουργούμε πλαίσια έτσι ώστε να υπάρχει κάποια δυνατότητα επανόρθωσης. Και έρχομαι σε αυτά που έλεγε ο σχετικά με την κάλυψη κατά 100%. Σε ορισμένε χώρε ισχύει ήδη το 100% και δεν πρέπει να τη ζητήσουμε να απομακρυνθούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε τα θέματα αυτά να τα ξαναθέσετε στα πλαίσια της γενικής ε, συζήτησης, ε, τότε ίσως εκεί κάποιοι να επικαλεστούν και την επικουρικότητα. για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έθεσε ο Σβέν σχετικά με το Solvency 2 δεν ξέρω αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια εκ νέου συζήτηση για το Solvency 2 πρέπει να περιμένουμε καταρχάς τις εκτελεστικές ρυθμίσεις οι οποίες προέρχονται από τον κανονισμό Solvency 2 η επάρκεια των κεφαλαίων, η δυνατότητα χρήσης του κεφαλαίου, ποια είναι τα ελάχιστα επίπεδα κεφαλαίου και ε, και πότε ο, ο, επόπτης, η εποπτική αρχή εμπλέκεται στη διαδικασία. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα επίπεδο ε, δυνατότητας ελέγχου και χρήσης ε, του Solvency 2 από την επιχείρηση μέσα σε μια συγκεκριμένη αγορά. Να δούμε λοιπόν τι υπάρχει διαθέσιμο σαν μέσο ελέγχου και από αυτά τα διαθέσιμα μέσα ποια είναι αυτά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα και όχι να αρχίσουμε να κάνουμε εκ νέου μία συζήτηση γύρω από το Solvency 2. Περιμένουμε την 1η Ιανουαρίου του 2013 έτσι και αλλιώς τις εκτελεστικές ρυθμίσεις και διευκρινήσεις για το Solvency 2. Ευχαριστώ Πίτα. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 12 το μεσημέρι στις 23 Μαρτίου, θα εξεταστούν στις 19 Απριλίου, θα ψηφιστούν στις 24 Μαΐου και στην δεύτερη Ολομέλεια του Ιουνίου θα ψηφιστούν. Περνάμε τώρα στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Γενική Οικονομική Διαχείριση, ο Γκούναρ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα διανύμω ένα σχέδιο της δομής της έκθεσης σε σχέση με τους γιώδες εισηγητές, σε σχέση με την προώθηση της συζήτησης πρωτού παρουσιαστεί η τελική έκθεση. Αλλά για να είμαι σύντομο και περιεκτικός, θα έλεγα πρώτα απ' όλα πρέπει να εξετάσουμε το γεγονός ότι η ισορροπία των παγκόσμιων οικονομιών, της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα είναι διαφορετική από στο παρελθόν. Τα περισσότερα παγκόσμια ιδρύματα <clears throat> περισσότερο σε σχέση μετά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τότε έγιναν πάρα πολλά πράγματα και με ταχύτητα τους ρυθμούς τα περισσότερα πράγματα άλλαξαν και σήμερα ζούμε σε μια τελείως διαφορετική οικονομική πραγματικότητα όπου η πιο δυναμική οικονομική ανάπτυξη συμβαίνει εκτός αυτού που ήταν η παγκόσμια οικονομία. Τότε όμως στο παρελθόν η παγκόσμια οικονομία ήταν η Δυτική Ευρώπη, η ίπα και κάποια άλλα μέρη του κόσμου επίσης. Αλλά αυτό είναι παρελθόν πλέον. Και αυτό ήταν τότε το κυρίαρχο μέρος στην οικονομία παγκόσμια. Σήμερα δεν συμβαίνουν όλα αυτά, βλέποντας τις αναδυόμενες οικονομίες των αναδυόμενων χωρών. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους ε, πίσω από την, την κρίση, την χρηματοοικονομική που είδαμε. Το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία δεν προσαρμόστηκε σε αυτές τις νέες ισορροπίες ε, που ε, έχουμε μπροστά μας και αντιμετωπίζουμε. Συζητώντας τις ισορροπίες και τις ανισορροπίες είναι σημαντικό πάντα να θυμόμαστε ότι πάντα υπήρχαν ανισορροπίες και αναντιστοιχίες επί δεκαετίες όταν βλέπαμε την φτώχεια στον τρίτο κόσμο να, να αυξάνεται και αυτό ήταν μέρος της ανισότητας χωρίς επενδύσεις και χωρίς ανάπτυξη σε τεράστια μέρη της παγκόσμιας οικονομίας και φτώχεια, ανέχεια τώρα αλλάζουν τα πράγματα και είναι σημαντικό πιστεύω ως ένα από τα σημεία, πολλά σημεία αφετηρίας και κίνησης. Κατά τα τελευταία 30 χρόνια είδαμε πάρα πολλούς σε παγκόσμια κλίμακα να ζουν σε σχετική ευημερία. Από ένα δις σε τέσσερα δις αυξήθηκαν και αυτό δημιουργεί τελείως διαφορετικούς όρους και διαφορετικές προϋποθέσεις για την παγκόσμια διακυβέρνηση και την παγκόσμια οικονομική τάξη πραγμάτων, αν μου επιτρέπετε η χρήση αυτού του όρου. Αυτό είναι που σημαντικό, είναι σημαντικό τώρα, είναι να πετύχουμε παγκόσμια θέματα και στόχους όπως διαφάνεια, θέματα όπως κανόνες και διατάξεις, σταθερότητα στο χρηματοοικονομικό δημοσιονομικό σύστημα. Πρέπει να κατανοήσουμε το τι γίνεται σε σχέση και με τα νομισματικά θέματα διότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά και στην επερχόμενη κρίση που είδαμε ότι επερχόταν, ήταν ότι οι διαφορετικές πολιτικές που είχαν υιοθετηθεί και οι ΙΠΑ είχαν ηγετικό ρόλο στο να δημιουργούν προβλήματα με την νομισματική πώληση που ακολουθούσαν. Και σήμερα ακόμα βλέποντας την νομισματική πολιτική των ΙΠΑ, βλέπουμε προβλήματα που δημιουργούνται νομισματικά στον υπόλοιπο κόσμο. Τα πράγματα είναι αλληλοσυνδεόμενα λοιπόν και εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Και όταν συζητάμε για ανισότητες πρέπει να θυμόμαστε ότι χρειάζονται δύο, όχι μόνο για να χορέψουν ταγκό, αλλά και δύο εμπλέκονται τουλάχιστον όσον αφορά την δημιουργία ανισοτήτων. Αυτό το θυμόμαστε όταν κάνουμε λόγο για πλεονάσματα και τα ε, συνεπαγόμενα προβλήματα. Επίσης όμως πρέπει να συζητούμε και τα προβλήματα των ελλημάτων. <clears throat> Διότι είναι τα ελλείμματα εκείνα τα οποία δημιουργούν ε, τα πλεονάσματα και ε, πολλές οικονομίες δαπανούσαν περισσότερα. Και αυτό ήταν ένα λόγο για πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν σε άλλε οικονομίε. Αν δεν κάνουμε λόγο για την Ευρώπη, τότε μπορούμε να δούμε τα άλλα τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας. Το πλεόνασμα βρίσκεται στην Κίνα βέβαια και είναι αποτέλεσμα των ελλημάτων στη ΣΥΠΑ αυτό το πλεόνασμα των Κινέζων. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα εξετάσουμε ταυτόχρονα αυτά τα δύο σκέλη. Πρέπει λοιπόν να στρέψουμε το βλέμμα προς το μέλλον με κάποια κέρια σημεία ως συμπεράσματα που πρέπει να συζητήσουμε ως θέματα, ως ζητήματα. Πρώτα απ' όλα τα παγκόσμια οικουμενικά θεσμικά όργανα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τέτοια παγκόσμια θεσμικά όργανα. Παράδειγμα, στο πλαίσιο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Η Λέσχη των 20, G20, πρέπει να διαδραματίσει ω ομάδα ένα σημαντικό ρόλο για τη διασφάλιση τη εφαρμογή και σεβασμού των κανόνων για τη διαφάνεια αλλά και για την ε, σταθερότητα. Κάνοντα λόγο, έχουμε κάνει πολλέ φορέ λόγο για θέματα σαν την ε, φερεγγιότητα και την ε, δυνατότητα ρευστότητα Solvency 2. Πράγματα, πράγμα που συνδέεται, για το, συνδέεται με το πώ αντιμετωπίζουμε τι ε, παγκόσμιες δομέ και τον συντονισμό του. Να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον, να δούμε ότι σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ω θεσμικό παγκόσμιο όργανο θα, πρέπει, θα έχει σημαντικό και έχει σημαντικό ρόλο και πρέπει να τεθούν υψηλέ προδιαγραφέ και απαιτήσει. Ακόμα και με την ομάδα ομάδα, την λέσχη των 20, G20 να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μείωση των ανισοτήτων, του πιο διαφορε... των ε, διαφορετικών τύπων που έχουμε. Και όταν συζητούμε τα θέματα ε, των νομισμάτων, το θέμα δεν είναι να έχουμε νέους κανόνες για την ανάπτυξη των νομισμάτων μας και τη μετεξέλιξή τους, αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα βασίζονται αυτά τα νομίσματα σε μια πιο κοντινή στην πραγματικότητα, οικονομική πραγματικότητα βάση. Καλό θα ήταν αυτό. Ταυτόχρονα όμως να λάβουμε υπόψη ότι και σχετική πειθαρχία θα απαιτείται για τις νομισματικές πολιτικές διότι η νομισματική πολιτική πολύ συχνά όπως είπα προκαλεί τα προβλήματα των διαφορετικών νομισμάτων. Και θα ήθελα να προσθέσω και ένα τρίτο στοιχείο σε όλο αυτό το σύνολο. Και αυτό είναι για να υπάρξει ισορροπία ή για να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και σταθεροποίηση στην παγκόσμια οικονομία πρέπει να δούμε και τι γίνεται, πώς λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Διότι το σημερινό παγκόσμιο εμπορικό σύστημα είναι ασυμμετρικό, μη συμμετρικό και δεν είναι επαρκώς ανοιχτές οι παγκόσμιες αγορές όπως θα έπρεπε να είναι. Και αυτό πάρα πολλές φορές αποβαίνει ε, προς, ε, ε, στην, με αρνητική επίπτωση βάρος του ευρώ. Και αυτό μπορεί μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη των ελλημάτων εκεί όπου υφίστανται αυτά τα ελλείμματα. Αν είχαμε ε, μια πολύ πιο ανοιχτή παγκόσμια ε, λειτουργία αυτού του συστήματο, αυτό θα ήταν επωφελέ και θα συνεισέφερε στην αύξηση των εξαγωγών και θα μείωνε τα ελλείμματα που έχουμε και ίσω θα δημιουργούσε και πλεονάσματα. Και πρέπει επίση, θα έλεγα, να λάβουμε υπόψη στη συνολική αυτή σφαιρική προσέγγιση, να λάβουμε υπόψη και τι γεωργικέ αγορέ. Διότι αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για πολλέ χώρε στον φτωχότερο κόσμο, του φτωχού κόσμου κόσμου να προωθήσουν τις εξαγωγές τους γεωργικών προϊόντων. Ξέρουμε πόσο ευαίσθητα είναι όλα αυτά τα θέματα και ποια σπουδαιότητα έχουν. Αν θέλουμε να καταλήξουμε όμως σε μια πιο ισόρροπη προσέγγιση της παγκόσμιας οικονομίας, ισορροπημένη προσέγγιση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας που σήμερα συνεισφέρουν σε αυτές τις ανισότητες και τις δυσαναλογίες. Στόχος μου είναι σε αυτή την έκθεση να προσπαθήσω και να καταφέρω αν γίνεται να θέσω ενώπιον μας τις κυριότερες ιδέες και στόχους, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε για την μεταξέλιξη των παγκόσμιων αυτών θεσμικών οργάνων, ώστε από το 2011 και εφ' να πορευθούμε προς αυτή την κατεύθυνση απέχοντας και παρεκκλίνοντας από τις παλαιότερες δομές και τις νοοτροπίες που είχαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε σχέση με την τότε νομισματική μεταρρύθμιση και τον κόσμο από τότε μέχρι σήμερα. Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων. Θα έχει όμως και σοβαρές επιπτώσεις, διότι αν μπορεί η Ευρώπη να αναπτύξει μια ε, ρεαλιστική προσέγγιση αυτών που μπορούμε να πετύχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και αν μπορέσει τότε να δημιουργήσει σταθερές δομές που θα είναι ε, ε, αντιπροσωπευτικές για την σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, τότε θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο για την μεταξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας στο μέλλον. Και μπορούμε να πούμε ότι βλέποντας τον σημερινό κόσμο, βλέποντας και τις εξελίξεις στην Ιαπωνία ακόμα σήμερα, χρειαζόμαστε απόλυτα σταθερά θεσμικά όργανα, παγκόσμια θεσμικά όργανα. Χρειαζόμαστε όμως και έναν πολιτικό στόχο που να εμπνέει αυτό το εγχείρημα. Ρεαλιστικά εγχειρήματα όχι μόνο λόγια, αλλά και στις πράξεις δημιουργώντας τα θεμέλια για αυτή τη μεταξέλιξη και πρόοδο. Προσβλέπω στη συζήτηση όχι μόνο εδώ, αλλά και μεταξύ και των σχεδόν εισηγητών και στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή όταν παρουσιάσω την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. On... Ευχαριστούμε, Κουνε. Δεν έχουμε εδώ πολλούς ε, σκιώδεις, αλλά πρώτα ο Ευχαριστώ. Η οικονομική κρίση ήταν ε, διεθνής κρίση ξεκίνησε από μία χώρα, αλλά βέβαια διαδόθηκε παντού. Η οικονομική κρίση ήταν και είναι διεθνής. Το θέμα του χρέους βρίσκεται και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και οι σφαιρικές ανισορροπίες, παγκόσμιες ανισορροπίες είναι παγκόσμιες. Τα διεθνή λοιπόν προβλήματα απαιτούν και παγκόσμιες λύσεις. Να θυμηθούμε ότι το Διεθνές ε, Νομισματικό Σύστημα κατέρευσε το 1971 και τώρα έχουμε μια προσωρινή λύση ουσιαστικά, από μια χρονιά στην άλλη. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα. Έχουμε αρκετό ρευστό και τι ποιότητα. Είναι σωστό να χρησιμοποιούμε εθνικά νομίσματα για να, πληρώσουμε, να κάνουμε διεθνείς πληρωμές. Συμφωνώ επίσης με το γεγονός ότι τα διεθνή, οι διεθνείς θεσμοί χρειάζονται. Το G20 είναι ένα ξεκίνημα. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε προς το μέλλον. Γιατί να μην ξεκινήσουμε να δούμε και κάτι άλλο. Μήπως πρέπει να θεσμοθετήσουμε μια διεθνή διακυβέρνηση με το G20 και να δούμε πώς συνδέεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους. Η Παγκόσμια Τράπεζα, FC, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κτλ. Είναι ίσως το χρειαζόμαστε πάντω μια διακυβέρνηση που το παρόν εξυπηρετείται από τους 20. Γίνονται όμως συζητήσει για να δούμε μήπως πρέπει να επισημοποιηθεί ακόμα περισσότερο, να θεσμοθετηθεί. Τα θέματα υπάρχουν. Διακυβέρνηση πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαφθοράς, να υπάρχει διαφάνεια. Υπάρχουν έπειτα τα νομισματικά ζητήματα. Υπάρχει ο πληθωρισμός που δημιουργείται εξαιτία ε, των τροφίμων ή του πετρελαίου ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό. Και άρα χρειαζόμαστε μια παγκόσμια σταθερότητα. Ως κοιόδης εισηγητής αναμένω τη συνεργασία μας με τον κύριο Χοκμαρ είναι ο εισηγητής και σίγουρα θα συνεργαστούμε καλά γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να συνεισφέρει. Ευχαριστούμε κυρία Χούμπνερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι Γκούναρ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά μπροστά σου. Ελπίζω να τα καταφέρεις και να μας δώσεις κάποιες ιδέες που να χρησιμοποιηθούν στην προσπάθεια επίλυση των προβλημάτων. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα και είναι αναπόσπαστο τμήμα της πραγματικότητας και του μέλλοντός μας. Η οικονομική διακυβέρνηση απαιτείται όχι μόνο γιατί σφαιρικά προβλήματα απαιτούν σφαιρικές λύσεις, παγκόσμια προβλήματα, παγκόσμιες λύσεις, αλλά οι παγκόσμιες αγορές έχουν ανάγκη από κανόνες. Οι διεθνείς αγορές είναι συνδυασμοί των εθνικών και γι' αυτό απαιτείται να υπάρχει μια κάποια ρύθμιση. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν μεγαλύτερη προσοχή στην διεθνή οικονομική διακυβέρνηση λόγω ακριβώς και των ανισοτήτων που διαπιστώνονται και θα πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις μόνο στην περίπτωση που ε, η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση είναι λειτουργική. Μέχρι τώρα έχουμε δει τι ανεπάρκειες υπάρχουν στον κόσμο, βλέπουμε τι μας λείπει, βλέπουμε ποια είναι τα κενά αρμοδιοτήτων που έχουν οι υπάρχοντες διεθνείς οργανισμοί. Αυτά όλα καλύπτονται από ανεπίσημες λύσεις οι οποίες ήρθαν στην επιφάνεια αρκετά γρήγορα όταν επήλθε η κρίση. Όλες αυτές, ε, όλες αυτές, όλοι αυτοί οι οργανισμοί ad hoc εξακολουθούν να λειτουργούν σήμερα λόγω ακριβώς της ανεπάρκειας των μόνιμων θεσμών της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό που έχει σημασία βέβαια σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης είναι η διαφάνεια και οι ad hoc αυτές οργανώσεις δεν μας δίνουν τη διαφάνεια η οποία απαιτείται και δεν είναι μόνιμη λύση για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε. Ο ρόλος αυτών των ανεπίσημων οργάνων σήμερα μας παρουσιάζεται επί τη βάση της, ε, των προτάσεων που προέρχονται από την ομάδα των 20 που αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Αν δει κανείς την ιστορία της ομάδας των 20 μπορεί να πει ότι έχει κάνει κάποια βήματα έτσι ώστε να χάσει η ομάδα των 7 ή των 8 τον ηγετικό ρόλο που είχε στο παρελθόν. Από την άλλη όμως, όταν βλέπει κανείς Εάν το G7 ή το G8 είναι σε θέση σήμερα να διεκδικήσει την ηγεσία θα έλεγα της διεθνούς οικονομικής διακυβέρνησης, νομίζω ότι δεν είναι κάτι τέτοιο σίγουρο. Γι' αυτό λοιπόν παρά την ύπαρξη και της ομάδας των 20 εξακολουθούμε να έχουμε μια σταθή κατάσταση σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης η οποία δεν θα πρέπει να διαχειριστεί να, δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί τα προβλήματα. Ήδη από το 2008 είχαμε τα πρώτα προβλήματα και ο συνδυασμός των διεθνών συμφερόντων δεν είναι εύκολος. Ένα τρίτο θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω και στο οποίο αναφέρθηκε ο Γκούναρ με άλλα λόγια είναι ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των συμμετεχόντων γιατί αλλιώς οι αποφάσεις δεν θα γίνουν ε, σεβαστές και δεν θα υπάρξουν μόνιμες λύσεις. Ε, το ερώτημά μου λοιπόν είναι και ελπίζω να δώσει απάντηση η έκθεσή σου. Είμαστε έτοιμοι άραγε σήμερα να έχουμε μια κοινή άποψη, ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Ή απλά θα πρέπει να φανούμε πραγματιστές και να μείνουμε εκεί όταν βλέπει τα διαφορετικά συμφέροντα, όταν βλέπει ε, τις ε, ε, αντισότητες οι οποίες υπάρχουν και τις αποκλίσεις μεταξύ των θέσεων των εθνικών κτλ. Όλα αυτά προκαλούνται από εθνικά φαινόμενα και από εθνικές διαδικασίες. Και δεν είμαι βέβαιος ότι σήμερα είμαστε σε θέση να έχουμε ακριβώς μια, ένα κοινό όραμα. και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ρεαλιστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γκούνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνοψίσουμε έτσι τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο για τη σημαντική συνεισφορά τους. Αυτό δείχνει ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. ότι έχει αλλάξει η οικονομία και γι' αυτό πήγαμε στους G20 από τους G7, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά, αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι σωστός αυτός ο τρόπος και έτσι συμμετέχουν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, γιατί με τους G7 βάλαμε τις μεγάλες οικονομίες επειδή ακριβώς είχαν μεγάλη σημασία, χωρίς να σημαίνει όμως ότι εκείνοι εκπροσωπούσαν και τα συμφέροντα ευρέως. Έπειτα, επηρεζόμαστε όλοι από την κρίση που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Όταν όμως συζητάμε για την ε, παγκόσμια οικονομία και τα παγκόσμια θεσμικά όργανα, πρέπει να μην ξεχνάμε και την παγκόσμια επιτυχία που είχαμε 30 χρόνια. από τότε δηλαδή που έχασαν την επιρροή τους στα μεγάλα θεσμικά όργανα στα μέσα του 80 που δεν είχαμε πια Bretton Woods που είχαμε εντελώς διαφορετικές παγκόσμιες δημοσιονομικές αγορές και από το ένα δις που ζούσε σε ευημερία στα 4-5 δις που ζουν σε ευημερία είναι μια σημαντική αλλαγή που πρέπει να την θυμόμαστε και να την στηρίζουμε. Μην την ξεχνάμε και στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν ένα παγκόσμιο πλαίσιο, διαφάνεια, ε, διαφερόμενες πλευρές. Όλα αυτά τα είπαν οι συνάδελφοι. Αλλά να υπάρχει και η ελαστικότητα, η ευελιξία για να μπορούμε να κινηθούμε. Είναι θέμα όρων, διότι θέλουμε μια ασταθερή κατάσταση, αλλά με ένα δυναμικό ανάπτυξης. Έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κούνερ. Όντω. η έκθεσή σου φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχουμε ιδιαίτερες προθεσμίες ακόμα, είναι χαλαρά τα πράγματα. Πάντως, θα παρουσιάσει το σχέδιό σου στις 19 Απριλίου. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι 10 Μαΐου. 14 Ιουνίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 19 Σεπτεμβρίου. Πράγμα που σημαίνει ότι στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Βλέπω εδώ όμως και το χρονοδιάγραμμα ε, του G20. Η τελευταία διάσκεψη είναι το Σεπτέμβριο, οπότε έχουμε βέβαια καιρό τον Οκτώβριο. Θεωρητικά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και 13, 14, 15 που έχει συνεδρίαση στο Παρίσι το FMSGP. Οπότε μήπως θα πρέπει να είναι στη δεύτερη του Οκτωβρίου. Δεν ξέρω. Σκέψου το. Για να προσαρμόσουμε ανάλογα το χρονοδιάγραμμα. Ναι, νομίζω ότι σωστό είναι αυτός ο στόχο. Γιατί όσο πιο γρήγορα έχουμε μια ατζέντα, μια μερίσια διάταξη γι' αυτό, τόσο το καλύτερο. Αλλά όντω έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μα ακόμα. Και ο σκιώδη ηγητή την ίδια γνώμη έχει. Καλώς. 19 Απριλίου έτσι κι αλλιώ είναι η επόμενη, ο επόμενος σταθμός στην διαδικασία αυτή. Έληξε η συνεδρίαση.